Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα στην αρχή της συνεδρίασης λοιπόν να καλωσορίσω τον Επίτροπο Γιωχάνες Χάν και θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όσους δεν έχω δει. Κάποιους από σας, σας έχω ήδη δει. Καλή χρονιά λοιπόν. Και να καλωσορίσω δύο νέα μέλη στην γραμματεία. Τη Βερόνικα Πατιχόβα, η οποία επέστρεψε μετά από μια μεγάλη απουσία και την κυρία Βετσέβα, η οποία είναι νέα συνάδελφος. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Σηκωθείτε για να σας δουν και οι συνάδελφοι. Σηκώστε το χέρι. Και να καλωσορίσουμε την Κριστίνα Τεγκέλντερε. Η ομάδα μας λοιπόν αυξάνεται σε πληθυσμό. Ελπίζω να κάνει τη δουλειά μας λίγο πιο εύκολη. Η γραμματεία πάντα έχει πάρα πολλή δουλειά και δύσκολη δουλειά, ανεξάρτητα από το ποιοι απαρτίζουν την Επιτροπή. Ελπίζω λοιπόν να δουλέψουμε λίγο πιο άνετα με τις νέες προστίκες. Μετά, ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη. Περνάμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει κάποια ερώτηση, σχόλιο, ε, αντίρρηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τότε θεωρείται εγκεκριμένη. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Υπάρχει διερμηνία σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των άλλων και στα ελληνικά. Τα πρακτικά της, ε, της συνεδρίασης της 4ης Δεκεμβρίου είναι στη διάθεσή σα, όπως επίσης και οι αποφάσεις των συντονιστών από τις 10 ε, Δεκεμβρίου. Υπάρχει σχόλιο? Όχι. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πώς είναι εγκεκριμένα. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έκθεση ε, με εισηγήτρια την υποφαινόμενη, απαλλαγή 2018, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι προσπάθησα να χτίσω γερά θεμέλια, μια σωστή βάση πάνω στην οποία θα μπορείτε εσείς να συνεισφέρετε μέσω των τροπολογιών σας. Η έκθεση λοιπόν αφορά την ετήσια απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προσπαθήσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε την ε, υπάρχουσα δομή του ελεκτικού συνεδρίου για να μην ε, μας κατηγορούν και ότι σε κάθε διαφορετική περίπτωση ακολουθούμε δική μας κατεύθυνση. Προσπαθήσαμε λοιπόν, ε, αφού εξετάσαμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, να κάνουμε τις δικές μας προσθήκες και τροποποιήσεις και να τονίσουμε τα σημεία που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο και σημαντικότερο θέμα για την έκθεση ήταν το κράτος δικαίου, έπειτα η χρηστή οικονομική διαχείριση, στη συνέχεια η αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων και σε αυτούς τους ε, τομείς κινήθηκαν οι τροπολογίες μας. Επίσης, στην ε, Ολομέλεια του ε, Δεκεμβρίου συζητήθηκε το θέμα της ε, Τσεχίας και το γεγονός ότι η, οικονομική δομή, τη διαχείριση της χώρας ε, χαρακτηρίζεται από ολιγαρχικά. Και δεν υπάρχει λοιπόν ε, δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή στα οικονομικά. Αυτό ήταν ένα προβληματικό σημείο. το οποίο σημείωσα και εγώ στην ε, δουλειά που έκανα κατά την κατάρτιση της έκθεσης. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει το θέμα αυτό. Υπάρχουν και θέματα ψηφιοποίηση αυτό, αυτή η ψηφιακή Ευρώπη που θέλουμε όλοι να έχουμε, που προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυστυχώ δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ψηφιακή πρόσβαση στην ε, πληροφορία και αυτό σημαίνει αύξηση ε, σημαντική της ε, γραφειοκρατίας. Θεωρούμε ότι η ψηφιοποίηση θα μειώσει το, τη γραφειοκρατία αλλά θα αυξήσει και την διαφάνεια. Θα αποφευθούν έτσι αρκετά προβλήματα. Γι' αυτό και ελπίζω να υπογράψουμε από κοινού μια τροπολογία έτσι ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της ψηφιοποίησης. Ελπίζω λοιπόν να έχω τη στήριξή σας αυτό. Έπειτα. Έχει προκύψει και το ερώτημα του ε, πόσα χρήματα θα πρέπει να δίδονται σε ένα μεμονωμένο άτομο. Στην ε, Επιτροπή Γεωργίας έχει συζητηθεί το θέμα εν ώψη του νέου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό βέβαια δεν ε, έχει σκοπό να αυξηθεί η γραφειοκρατία, αλλά το αντίθετο. Έχουμε συζητήσει λοιπόν ε, με τους συνάδελφους και τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας. Έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό από κοινού. Θα συζητήσουμε και με τους ε, υπεύθυνου στην Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο και Οικονομικών έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Επίσης, μας απασχόλησε και το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος ε, στην Γεωργία, στην Ιταλία. Όπως επίσης και θέματα διαφάνειας. Εδώ έχουμε παρατηρήσει πως υπάρχουν πολλοί τομείς που επιδέχονται βελτίωσης. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε την ανάγκη για βελτίωση. Επίσης, καλωσορίζουμε την ε, πρόθεση του ελεκτικού συνεδρίου να ε, διευρύνει λίγο τον, ε, το σύστημα διεξαγωγής ελέγχων, τη διεξαγωγή ελέγχων από ανεξάρτητες εθνικές αρχές. Έπειτα, ασχοληθήκαμε και με το θέμα του ελέγχου επιδόσεων, performance audit, ε, τον ορισμό του. Τι σημαίνει δηλαδή ο έλεγχος επιδόσεων. Χρειάζεται να συλλέξουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε έναν πλήρη ορισμό. Έπειτα, φορολογική απάτη, τελωνιακή απάτη. Εδώ χρειάζεται ενίσχυση των τελωνιακών αρχών για την καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να καταθέσουμε σχετική τροπολογία για το θέμα αυτό. Μετά, γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων στον ε, χώρο της επιστήμης και της ε, επιστημονικής έρευνας, αριστεία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φυσικά και θέλουμε αριστεία, όμως ε, πρέπει να ασχοληθούμε με την γεωγραφική κατανομή της αριστείας και να φροντίσουμε έτσι ώστε όλα τα ε, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποφελούνται από χρηματοδότηση. Εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η έρευνα σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και να έρθει πιο ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων, κάτι που δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Έπειτα έχουμε και τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, διάφορες εκκρεμότητες ε, από το προηγούμενο έτος. Αυτό μας έχει απασχολήσει και άλλες φορές. Και προσπαθούμε μέσω της έκθεσής μας να πιέσουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να καθαριστούν αυτοί οι λογαριασμοί. Χρησιμοποιώντας και τη μέθοδο νήσιν 3. Έρχεται ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών και ελπίζουμε λοιπόν να έχουν λυθεί αυτές οι κρεμότητες μέχρι τότε. Έπειτα, κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχει ανάγκη για δίκαιη κατανομή της ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Εδώ έχουμε κάνει δικές μας προσθήκες. Έπειτα ασχολούμαστε με το μηχανισμό κατανομής χρηματοδότησης στους αγρότες. Χρειάζεται συμπερίληψη και των ε, εθνικών αρχών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα προσφυγής των δικαιωχών στις εθνικές αρχές, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι, έχει γίνει κάποια, ότι έχουν αδικηθεί, έχει γίνει κάποια παρατυπία. Έπειτα ασχολούμαστε με την αναποτελεσματικότητα του πρασινίσματος. Είναι κάτι που έχει τονίσει στην έκθεσή του το ελεκτικό συνέδριο στο πλαίσιο της νέας πράσινης συμφωνίας θα πρέπει να ε, ζητήσουμε αποτελεσματικές ε, μεθόδους πρασινίσματος χωρίς πολλή γραφειοκρατία. Και επίσης ζητούμε βελτίωση των ε, υποδομών της ε, βιομηχανίας ε, και ε, της γεωργικής βιομηχανίας έτσι ώστε και οι μικροί αγρότες να μπορέσουν να επωφεληθούν. Έπειτα ασχολούμαστε με τα hot spot. Θέλουμε βελτίωση των υποδομών ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία και κάποιες άλλες χώρες κυρίως για τα παιδιά που φιλοξενούνται στις υποδομές αυτές. Ασχολούμαστε και με το φαινόμενο της κατάχρησης κονδυλίων και με το θέμα της ε, διαφάνειας και της λογοδοσίας στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Έχουμε συνομιλήσει με τους συναδέλφους ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι ότι το κράτος της Ερυθρέας χρησιμοποιεί την διεθνή βοήθεια για να προωθήσει ε, να προωθήσει τη δουλεία. Αυτά είναι δημοσιευμένα ήδη στο διεθνή τύπο, στους New York Times. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που οι New York Times έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα αυτό και τα θέματα της χρηματοδότησης. Ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Έχουμε, έχουμε ζητήσει απαντήσεις από τον Επίτροπο Μίμητσα, μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση. Ο... Ο ΙΕ βέβαια πρέπει να λογοδοτήσει διότι σε τελική ανάλυση χρησιμοποιούνται και δικά μα κονδύλια στην ε, Ερυθρέα. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια επίσημη, ένα επίσημο ερώτημα προς την κυβέρνηση της ε, χώρας, διότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση πληροφοριών που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για να μπορέσουμε να κρίνουμε την κατάσταση. Αναφέρεται λοιπόν στην απαλλαγή μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης το θέμα αυτό. Η συνεργασία δηλαδή με τις τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανάπτυξης. Επίσης έχουν γίνει ορισμένες ε, διορθώσεις γλωσσικού τύπου και προσπάθησα να σας δώσω μια πολύ συνοπτική εικόνα λοιπόν ε, ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης. Ε, θα κατατεθούν τροπολογίες για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι πράσινοι έχουν καταθέσει τροπολογίες και έχουν δείξει μεγάλη ευαισθησία απέναντι στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ωστόσο είναι κάτι που πρέπει να σημειωθεί. Έχει αναφερθεί και το παράδειγμα μιας τουρκικής μη κυβερνητικής οργάνωσης. Κάθε φορά που τίθεται θέμα διαφάνειας ε, είναι ένα θέμα που είναι μεν δεκτό όταν πρόκειται για κράτη-μέλη, αλλά όχι όταν πρόκειται για μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ε, δεν γίνεται όμως έτσι να υπάρχει μια προτιμησιακή συμπεριφορά. Δεν μπορούν να μας λένε να μην αγγίζουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Χρειάζεται όλοι, λοιπόν, να διέπονται από ίσους όρους, να υπάρχει ένα μητρό διαφάνειας για να ξέρουμε ποιος έχει πάρει τι και πώς το έχει χρησιμοποιήσει, να υπάρχει λογοδοσία. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να υπενθυμίσω πως έχω καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε έτσι ώστε να έχουμε μια καλή έκθεση η οποία θα βοηθήσει την Κομισιόν. Αυτά από μένα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Πένκοβα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους που δεν έχω δει ακόμη Καλή χρονιά. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την παρουσίαση και για την έκθεση. Θεωρούμε πως καλύπτει τις περισσότερες πτυχές, τα περισσότερα ζητήματα που έχουμε συστήσει και τους τελευταίους μήνες με το ελεγκτικό συνέδριο και στις ακροάσεις που είχαμε με τους επιτρόπους εδώ στην Επιτροπή μας. Βεβαίως και θεωρούμε θετικό το ότι επισημαίνεται τα βασικά ζητήματα που άπτονται τη επίδοση, των επιδόσεων και όχι των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. Όπως λέει και το ελεγκτικό, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων για την έρευνα. Το σημειώνουμε και αυτό. Είναι σημαντικό επίσης ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πορισμάτων των ελέγχων του ελεγκτικού ε, και της Κομισιόν και πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση της μεθοδολογίας της Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές στις συζητήσεις ε, με τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή μας το έχουμε θέσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, θα επεξεργαστούμε τις τροπολογίες μας και θα σας πω τι θέλουμε να περιληφθεί. Είπα ήδη ότι τα βασικότερα καλύπτονται, αλλά θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη Ε, προσοχή στην άμεση, έμεση και συνδιαχείριση στις τρεις αυτές πτυχές. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Θέλουμε επίσης να περιληφθεί σε επιδόσεις και η βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή, μάλλον στην ε, εκτέλεση των στόχων και των αναπτυξιακών. Να δούμε τι γίνεται με τη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών που δυσκολεύονταν από κονδύλια και πώς αυτή η προχωρήσει. Η Κομισιόν νομίζουμε ότι θα πρέπει να παρέχει βοήθεια στα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή και ιδίω στα μέτρα καταπολέμηση απάτης για καλύτερε επιδόσει. Με εστίαση στι και στο ΕΤΠΑ κυρίω. Φυσικά θέλουμε το μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθορά απάτης, στους συγκρούσεις συμφερόντων, πάτε και να το ε, ενισχύσουμε. Τα βασικά αυτά είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και την καλή μέχρι τώρα δουλειά. Και όπως είπα ήδη είναι αρκετά αναλυτική έκθεση, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολιβιέ Σαστέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω γαλλικά, όπως καταλάβατε. Και εγώ θέλω να σας ε, ευχηθώ ευτυχισμένο τον έτος ε, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, και σε όλους τους συνεργάτες μας. Θα μας βοηθήσουν ε, αυτή τη χρονιά το 2020 και θέλω καταρχήν να σας ε, συγχαρώ εσάς κύριε Πρόεδρε για τη δουλειά σας ε, και ως εισηγήτρια λάβατε εδώ υπόψη όλα όσα έχουμε ακούσει, όλα όσα έχουμε συζητήσει στις διάφορες μας ε, συνεδριάσεις με την Επιτροπή και με το Ελεγκτικό Συνέδριο και στις συνεδριάσεις μεταξύ μας. Έχετε λοιπόν συμπεριλάβει ήδη στην έκθεσή σας πολλές παρατηρήσεις, πολλές προτεραιότητες και ιδίως αυτές τις οποίες και εμείς είχαμε αναδείξει ως ομάδα. Επίσης συμφωνώ πολύ με την εισαγωγική σας παρέμβαση και κάποιες συμπληρωματικές ε, παρατηρήσεις ε, που είπατε ότι θέλετε να περιλάβετε, όπως και κάποιες επιπλέον τροπολογίες που θέλετε να καταθέσετε. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για την ε, έγκριση της έκθεσης. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα σημεία. Εστίαση μεγάλη δίνεται στους δείκτες επιδόσεων και αυτό είναι σημαντικό κατ' διότι είναι και ο σκελετός της δράσης μας, ε, είναι η βάση της δουλειάς που κάνουμε πρέπει να επενδύσουμε σε πολιτικές που λειτουργούν και όχι σε αυτές που αντιβαίνουν και στην κοινή οικονομική λογική. Βλέπουμε επίσης ότι ε, υπάρχει ε, προ... δεν υπάρχει ισχυρό μεγάλο πρόβλημα πλέον με τα ποσοστά ασφάλματος, αλλά πρέπει να δούμε το ποιοτικό στοιχείο. Θα δούμε και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, γιατί ζητείται ευθυγράμμιση της Κομισιόν με τη μεθοδολογία του ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά τα ασφάλματα και αυτό είναι θετικό. Αναφέρεται επίσης ορισμένε εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου στην εκθέσή σας και θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μία έτσι πιο τεταμένη παράγραφο που θα αναφέρεται ακριβώς ε, στο έργο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Είμαι λίγο επιφυλακτικός για το να δοθεί προβολή, τέλο πάντων να φερθούν συγκεκριμένα κάποιε χώρε ε, στο πλαίσιο προβληματική που αναφέρατε. Εγώ θα έλεγα να έχουμε μια πιο γενική προσέγγιση. Είναι νομίζω πιο ενδεδειγμένο αυτό από το name and shame το να, επωνομάζουμε, να κατονομάζουμε και να επωνυδίζουμε ορισμένους. Σε ό,τι δεν αφορά τις τροπολογίες και εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για την κατάρριξη και πολλαπλασιασμό των ειδών ε, τύπου σφάλματος ε, ε σε ό,τι αφορά το κλείσιμο, υπολοιματικό κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε ώστε να έχουμε, το είπα και πριν, μία και μόνη μεθοδολογία. Επίση, πρέπει να γίνουν και προσπάθειε, θα έλεγα, παιδαγωγικού χαρακτήρα προ την Κομισιόν ότι αφορά την πολυπλοκότητα των κανόνων. Διότι όσο πιο πολύπλοκη, τόσο μεγαλύτερο και το ποσοστό σφάλματο. Οι εθνικέ περιφερειακέ διοικήσει Επίσης πρέπει να πλαισιωθούν καλύτερα, να υπάρχει μια παρακολούθηση, τεχνική βοήθεια, πληροφόρηση, σεμινάρια για να υπάρξει και μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφηση σε μερικά κράτη-μέλη που ναι, μεν έχουν μέσα, αλλά ε, στερούνται ενίοτε ε, των οικονομικών, ανθρώπινων, διοικητικών ε, πόρων και αυτό σίγουρα συνιστά μεγάλη απώλεια σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Επίσης, επιστέγνωσμα όλων αυτών είναι η διοικητική απλούστευση, το είπατε και εσείς. Και φυσικά έρχεται να κλείσει και τα δύο πρώτα σημεία μου ω συμπέρασμα. Πρέπει η διοικητική απλούστευση να είναι στο επίκεντρο και των στόχων της Κομισιόν, διότι αν υπάρχει διοικητική πολυπλοκότητα, αυξάνονται τα ποσοστά σφάλματος, ιδίως για το μη επιλέξιμο κόστος και βέβαια έχει και αποτρεπτικό αποτέλεσμα απέναντι σε μικρές δομές και δι απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γίνονται προσπάθειες σε κάποιους τομείς, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και σε άλλους. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πούμε πως ο δικός μας ο ρόλος είναι να ελέγχουμε την χρηστή εκτέλεση των ε, λογαριασμών και όχι να παρεμβαίνουμε στις ε, τομείς αρμοδιότητας άλλων επιτροπών όπως είναι η Άγκρη ή η η Και να συγχαρώ το ελεκτικό συνέδριο, το είπα και το επαναλαμβάνω, ότι πραγματικά μας βοηθούν, μας δίνουν τροφή για συζήτηση για προβληματισμό θα πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο τις ειδικέ εκθέσεις και τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Γίνεται στην έκθεσή σας για την απαλλαγή μηνίας ορισμένες εκθέσεις όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τη ΦΠΑ. Πραγματικά φαντάζομαι ότι για τις ε, συζητήσεις επί του προπολογισμού έχετε ε, ξενυχτήσει κυρία Πρόεδρε για να κερδίσουμε κάποια χρήματα, εκατομμύρια ίσως και βλέπουμε δισεκατομμύρια να φεύγουν από τα χέρια μας ε, λόγω της μη καλής εκτέλεσης και, της, και στην περίπτωση των τελωνιακών. Κάτι το οποίο δεν έχει νομίζω επισημανθεί στο σημείο που εγώ θα ήθελα είναι η ψηφιοποίηση. Πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων, όπως έχει γίνει παραδείγματος χάρη με τις άμεσες ενισχύσεις, ε, άμεσες πληρωμές στη γεωργία, στην κοινή γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και την διάσταση του φύλου στην έκθεση. Να μπορούμε να ποσοτικοποιούμε ε, τι γίνεται με τα ερευνητικά προγράμματα ε, ότι πρέπει δηλαδή να υπάρχει ισομερής κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτά έχω να πω σε σχέση με το σχέδιο έκτη. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βιόλα Φονκράμ. Κράμ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να σας συγχαρώ και εγώ και να ευχηθώ καλή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μόνικα Χολμάρ για το πρώτο αυτό σχέδιο Πράγματι, ε, έχουμε δουλειά, θα δούμε και τις νέες τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι είναι καλό να ε, λάβουμε υπόψη μας κάτι το οποίο λέει και το ελεγκτικό συνέδριο. Ότι δηλαδή σε ορισμένα κράτη-μέλη φαίνεται να υπάρχουν συστηματικές αδυναμίες, όπως μεταξύ άλλων στις δειγματολογικές αυτές έρευνες που γίνονται και πώς ανακαλύπτονται ε, ή διαπιστώνονται οι παρατυπίες και τα διάφορα προβλήματα. Επίσης, ε, νομίζω ότι και από πολιτικής ε, πλευράς υπάρχουν αυτοί οι στόχοι. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον κάτι ανάλογο. Θα πρέπει να δούμε όταν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους εκτελεστικούς οργανισμούς ή τους επιθεωρητές στα κράτη-μέλη. Ε, σε σχέση δηλαδή με το πώς αξιοποιούνται οι πόροι, αν γίνεται κατάχρηση ή όχι. Και κάτι που ε, το λέμε πολλές φορές και έρχομαι στον τομέα της γεωργίας, πρόσφατα ακούσαμε κάποιες ε, πολιτικές προσωπικότητες να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά εγώ επανέρχομαι στο ότι Υπήρξαν πολλές εκθέσεις και αναφορές από την Κομισιόν προ την Όλαφ και η Όλαφ ερεύνησε τις σχετικέ υποθέσεις όπου γίνεται λόγο για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα έτη από 2012-2018 έχουμε 208 υποθέσεις ε, ε, που, για τις οποίες έκανε συστάσεις η Όλαφ και μερώθηκαν εθνικές αρχές. Αλλά τελικά φαίνεται να μην έχει συμβεί τίποτε. Και αυτό σημαίνει ότι σε πολλά άλλα συγκεκριμένα κράτη-μέλη δεν ε, υπάρχει ενδιαφέρον να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, τα συστηματικά κρούσματα απάτης και όταν ε, τα πράγματα είναι τόσο εξόφθαλμα και όταν και η Κομισιόν και η Όλαφ δεν μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο, θα πρέπει οι αρχές, που είναι πολύ σημαντικές για όλους μας, και τις αναφέρουμε συνέχεια, όταν πρόκειται για κράτη-μέλη διεφθαρμένα, όταν πρόκειται για κρούσματα διαφθόρας, τότε θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει μέσα στο παιχνίδι. Είναι καλό που υπάρχει αυτό το γραφείο, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ε, και θέλω να το πω δημοσία για μια ακόμη φορά ότι η εισαγγελία ε, ουσιαστικά πλήττεται από χρόνια υποχρηματοδότηση. και τα υποθέσεις ε, με τις οποίες αστικά κατακλίζονται είναι τριπλάσιες, τετραπλάσιες ε, και έχουμε την Όλαφ που δεν μπορεί να ερευνήσει περαιτέρω κάποιες υποθέσεις. Η εισαγγελία δεν είναι στελεχωμένη επαρκώς, οπότε ούτε το 2020 η υπερκοδότηση που προβλέπεται, ούτε με το πι θα καλυφθεί το πρόβλημα και αυτό είναι μείζον ζήτημα αξιοπιστίας. Είναι πλήγμα για την αξιοπιστία μας, για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί που γίνεται η αντιμετώπιση της διαφθοράς, ε, η κοινωνία μας ε, απογοητεύεται, βλέπει ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. και θα πρέπει να υπάρχει και μια κατάλληλη δικασία ε, να ε, επιλύονται αυτές οι υποθέσεις και σε επίπεδο εισαγγελία. Είναι πιθανό τελικά να υπάρξει αποτυχία. Και είναι μεγάλες οι πιθανότητες ε, για κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να επεξεργαστούμε αυτό το θέμα πάρα πολύ και κατεπηγόντως ανέφερε και κάποια άλλα θέματα η Μόνικα Χολμάγερ. Μιλήσαμε για το λόγο land grabbing στην πολιτική γεωργία των αρπαγηγιών που είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από τη ρίζα του και μπορεί να έχουμε αυτό το 37,5% ε, των ενισχύσεων των γικών. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε τι κίνητρα είναι λογικά ε, πέραν του τι ισχύει τώρα. Ε, τι διαφορετικά θα μπορούσε να γίνει δηλαδή στον τομέα αυτό. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει. Και οι συμβάσεις και συμφωνίες που μας επιβάλλουν να χρηματοδοτήσουμε κάποιους στόχους και κάποιες πολιτικές. Δεν κάνουν λόγο για ε, εξασφάλιση του δήματο. Αλλά λόγο για αύξηση τη παραγωγικότητα, για σταθεροποίηση των αγορών, για ενεργειακή ασφα... μάλλον ασφάλεια του εφοδιασμού κτλ. Δηλαδή, εκεί στηριζόμαστε, στη διάθεση κονδυλίων για την αύξηση της παραγωγικότητας. Όμω η κοινωνική πολιτική που βρίσκεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να το ακούσει αυτό, αλλά εγώ θέλω να σα το υπενθυμίσω. Όταν έχουμε γεωργική μεταρρύθμιση που θέλει να είναι άξια του ονόματος, θα πρέπει να τα δούμε αλλιώς τα πράγματα. Για να αντιμετωπίσουμε την ε, τον ενδυμικό πειρασμό, αν θέλετε, για διαφθορά στη γεωργία. Θετικά λοιπόν αυτά που είπες Μόνικα και σε σχέση με το τελικά ποιος είναι ο δικαιούχος ωφελείται από τις γιορκές επιδοτήσεις. Πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τη σώρευση κεφαλαίου. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται κατεπηγόντως είναι περισσότερη διαφάνεια σε αφορά την διοκτησία της γης. Πού πηγαίνουν τα χρήματα και νομίζω ότι στην Επιτροπή μας υπάρχει η μεγάλη βούληση να το δούμε σε βάθος Είπε και εσύ ότι υπάρχουν και άλλε επιτροπέ που θα συμμετέχουν, τι ανέφερε και είναι καλό ε, στοχευμένα να το αντιμετωπίσουν το θέμα και ε, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συνομιλήσουμε με κάποια κράτη-μέλη συγκεκριμένα. Αυτό θα κάνει καλό στην αξιοπιστία των θεσμών. Ε, εν παρόδο, το είπε και ο Σναυστορινιού, να αναφέρω και εγώ το θέμα της επιστήμης. Πολύ σημαντικό να μην μιλάμε μόνο για την ε, επιτυχία στις επιστήμες. Υπάρχουν επενδύσεις και στο γεωργικό τομέα. Μπορεί να αποδώσουν μετά από 5, 10, 20 χρόνια. Τότε να αποσβεθούν. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην βάζουμε ε, τόση, ε, να μην δίνουμε τόση σημασία στην βραχυπρόθεσμη μέτρηση ε, των επιδόσεων, του output. ή να μην κεντρωθούμε τόσο στο λεγόμενο success στις επιτυχίες ή να δώσουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ιδίως για το επιστημονικό έργο. Κάτι που το βλέπουμε είναι κριτικό μάτι είναι η συνεργασία με τρίτες χώρες, Κίνα, ε, και τη Huawei. Το αναφέρω συγκεκριμένα και είναι και εδώ ο τα ακούει όλα αυτά. Ε, θέλουμε ανταλλαγή σίγουρα δεδομένων σε αυτόν τον ευρύ επιστημονικό χώρο, αλλά ε, τη Huawei ε, στο, στην έκθεσή σου την κατονομάζεις, ε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα εμείς πώς ε, αντιλαμβανόμαστε τη συνεργασία μας με αυτόν τον παγκόσμιο πρωταγωνιστή και πώς θα θέλαμε να είναι Υπάρχουν και στρατηγικές επιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις υποτιμήσουμε. Συνολικά και το λες και αυτό, ε, ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω από την Κομισιόν, να είναι κάτι πιο ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά το καθαρό κέρδος ε, των ε, πολιτών από τις ταπάνες η γεωργική πολιτική εδώ ακόμα. Ε, παρουσιάσει πολλά ελλείμματα, ε, είτε ε, στην κτηνοτροφία, είτε στη βιοπικιλότητα, στιγματική αλλαγή και πραγματικά ουσιαστικά υπάρχει σπατάληση διασπάθηση το 1% των πόρων που διατέθονται για όλα αυτά. Τα λένε και οι επιστημονικοί οργανισμοί αρμόδιοι, τα λέει και το ελεγκτικό συνέδριο και σε σχέση με τη νέα μεταρρύθμιση της Κομισιόν, ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε σε αυτήν όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, όπως είπες, θα πρέπει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα όχι απλά για την ε, δήλωση κάποιων και την ε, δημοσιοποιήσει κάποιο περιστατικό, αλλά και μία, ένα πρόγραμμα προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντο. Και η ανωνυμία πρέπει να προστατεύεται στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορε γλώσσε. Ε, θα πρέπει να οργανωθούν όλα αυτά για να υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση, πληροφόρηση. Και τέλος, μίλησες για τον έλεγχο των ΜΚΟ, ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μια περίπτωση ε, που πήγαν εκεί κάποια χρήματα. Ναι, εγώ συμφωνώ να υπάρχει διαφάνεια ε, και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ότι είναι ένα στόχος αυτός ε, ο έλεγχος των ΜΚΟ, αλλά ίσως κάποιες φορές υπάρχουν άλλοι στόχοι και άλλα κίνητρα από πίσω. μην ε, υπερφορτώσουμε με κριτήρια, ε, υποχρεώσεις ε, και ανάγκη δημοσιοποίηση λοιπά της πολύ μικρές ΜΚΟ. Το ξέρω από την προηγούμενη μου δραστηριότητα. Ουκρανία, συνεργασία. Ουσιαστικά ποτέ δεν κατέφτανε αίτηση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πολύ μικρές ΜΚΟ, γιατί ξέρω δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα και με αυτό το Ίδρυμα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Ε, αλλά αυτή η γενική προσέγγιση ε, σε ό,τι αφορά τις ΜΚΟ μας ε, δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον, στο ECR. Ο κύριος Τσαρνέτσκι δεν είναι εδώ. Θα ήθελε κάποιος να μιλήσει στη θέση του. Δεν βλέπω κάποιον. Ο κύριος Φλάναγκαν επίσης λείπει. Από την κούε θα ήθελε κάποιο το λόγο. Όχι. Τότε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χάν για να κάνει κάποια σχόλια στα όσα άκουσαμε μέχρι τώρα. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς ως εισηγήτρια για αυτήν την ε, έκθεση, αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ε, αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους πάρα πολύ σημαντικά θέματα και ως ε, πρώην υπουργό για επιστημονικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να τονίσω ότι πρέπει να προωθείται και να προάγεται η επιστημονική έρευνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειάζονται επενδύσει ε, και με την ιδιότητά μου ως Επίτροπος για Περιφερειακά Ζητήματα προσπάθησα να βάλω την επιστήμη πολύ ψηλά στη λίστα των ε, προτεραιοτήτων της περιφερειακής ανάπτυξης. Χρειάζεται όμως από τη μία να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, ιδιαίτερα στις πρώην κομμουνιστικές ε, χώρες, όπου παραδοσιακά οι επιστημονική έρευνα λάμβανε χώρα στα πανεπιστήμια, στα ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολλές φορές ε, παρατηρούνταν ελλείψεις ε, σε επιστημονικό προσωπικό. Αυτό το είδαμε και σε πολύ γνωστά πανεπιστήμια όπως το Χούμπολ του, του Βερολίνου. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να βελτιωθούν αυτές οι υποδομές. Σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, στην Πράγα, ε, είναι προφανής η κατάσταση. Ε, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, όμως ε, το θα μπορούσε να αποκεντρωθεί η εκπαίδευση επίσης. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ε, επιχορηγήσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσουμε με λεπτομέρειες ποιοι λαμβάνουν, ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτών των ε, επιχορηγήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο δίκαιη κατανομή γεωγραφικά. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ε, διαρροή εγκεφάλων. Έχω ε, ο ίδιος προσωπική εμπειρία, έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ε, επιστήμονες οι οποίοι έχουν φύγει από τις χώρες τους για να κάνουν το ερευνητικό τους έργο σε πανεπιστήμια με καλύτερες υποδομές και μου είπαν ότι θα προτιμούσαν, θα, θα, γύριζαν πίσω εάν υπήρχαν οι κατάλληλε προϋποθέσεις γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να διαφυλάξουμε αυτές, ε, αυτή την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα μυαλά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να ριστέψουμε στην Ευρώπη. Ε, θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαι συναισθηματικός ε, για αυτό που λέω, όμως υπάρχει και οικονομική διάσταση σε αυτό, οικονομική ανάπτυξη που θα συνοδεύσει το ερευνητικό έργο. Το τονίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν υποδομές ε, και υλικοτεχνικές, να γίνουν βελτιώσεις και η αριστεία θα πρέπει να παραμείνει κριτήριο χρηματοδότησης. Ε. Και εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όμως ε, γεωγραφικά ε, κριτήρια και οι διαφορές που υπάρχουν από κράτος σε κράτος. Επίσης, ε, αναφέρθηκε και το θέμα της ε, συλλογής πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συλλογής Στοιχείων. Εδώ θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να μοιράζονται την πληροφορία, να υπάρχει πρόσβαση σε όλους. Θα πρέπει και εδώ να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για τη διαλειτουργικότητα. Και για να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για εκείνους που τα ζητούν και β για να υπάρξει κάποιο μητρό το οποίο θα είναι προσβάσιμο και ηλεκτρονικά. Ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε θαύματα και να δημιουργήσουμε νέο software για να γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες ε, υποδομές έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Νομίζω πως αν βελτιωθεί η πρόσβαση θα μπορέσουμε εκ των προτέρων να αποφύγουμε πολλά προβλήματα και να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Σε σχέση με αυτό, να πω δύο λόγια και για την απλούστευση που αναφέρεται στην ε, έκθεση σε όλους τους τομείς χρειάζεται αυτή η απλούστευση. και θα σταθώ στη χώρα που γνωρίζω περισσότερο από όλες, τη δική μου δηλαδή, την Αυστρία, και εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, υπάρχει υπερθεματισμό σε ό,τι αφορά την ε, χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να φαίνεται, θα πρέπει να υπάρχει κάποια καταγραφή σε ένα μητρό, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι πού ε, πηγαίνουν τα χρήματα. Αυτή η γραφειοκρατία είναι πραγματικό όνειδος για πολλές χώρες. Μετά, αναφερθήκατε στον ορισμό των επιδόσεων. Πώς μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε τις ε, επιδόσεις Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και κάποιο καιρό με το ελεκτικό συνέδριο, με τους ελεκτές. Ε, συζητιέται το ενδεχόμενο να υπάρξει μια πολιτική αξιολόγηση και συνοδευτικά μέτρα. Τα κράτη-μέλη εξάλλου θα είναι εκείνα που θα πρέπει να εκτελέσουν τις ε, οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Στηρίζω λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο στην προσπάθειά του να βελτιώσει τους ελέγχους επιδόσεων. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους παραδοσιακούς ίδιους πόρους έτσι ώστε να, αποφεύγονται, να ανακαλύπτονται και να αποφεύγονται οι περιπτώσεις κατάχρησης. Διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των συνθήκων σε ορισμένα κράτη-μέλη, όμως χρειάζεται συνεργασία αμφίδρομη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή ε, την ε, ψηφιακή την βελτίωση της ψηφιοποίησης, ψηφιακή διασύνδεση, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Ε, και παρεμπιπτόντως αυτό πρέπει να συνδεθεί και με το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, αν πάμε από τον νησιν στο νη συν 2, αν γυρίσουμε πίσω δηλαδή, τότε θα αλλάξουν πάρα πολλά. Οι βασικές, οι βασικές όμως, ε, το, το ζητούμενο μάλλον είναι να μην καθυστερήσει το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάθε καθυστέρηση κοστίζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, νομίζω πως ήδη υπόθηκαν όλα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα λέτε. Είναι εκ των όνου, φαν, εκ των προϋπόθεση διαφάνεια. Γι' αυτό και χρειάζεται σωστή νομοθεσία. Τώρα, από την εμπειρία μου ως ε, Επίτροπος για Περιφερειακά Ζητήματα, θεωρώ πως ε, θα πως θα μπορούσαμε και θα ήταν σωστό να υπάρχει αυτό το naming and shaming, να κατονομάζουμε τις ε, περιπτώσεις που θα πρέπει να μπουν σε μια μαύρη λίστα εντό εισαγωγικών, έτσι ώστε να λειτουργούν ως παραδείγματα προς αποφυγή. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, υπάρχουν αυτές οι διστάρετες περιπτώσεις και θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Τώρα, το που άκουσα για τους ενιαίους ελέγχους είναι μεν επιθυμητό. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και για ψηφιακή διαδικασία, ψηφιακούς ελέγχους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντομεύσουμε το έργο των ελεκτών. Αυτά προς το παρόν από μένα. Ε, να πω επίσης για τη σύγκρουση συμφερόντων ότι έχουμε συζητήσει και το Δεκέμβριο και έχουμε δει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε λύση. Θα Πρέπει φυσικά να ακούσουμε και τι μας λέει το ένστικτό μας ότι είναι σίγουρα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτήν την ολιγαρχική δομή η οποία φυσικά δεν ωφελεί πουθενά και παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις. Και σίγουρα αυτές οι ολιγαρχικές δομές όπου παρεμβαίνουν υπέρ το δέον ε, στο έργο της ε, διακυβέρνησης μιας χώρας δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Αυτά από μένα σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ να πω κι εγώ κάτι πάνω στην έκθεση. Νομίζω πως δεν θα σταματήσουμε τη συζήτηση, δεν θα έχει τέλος ε, αν ανοίξουμε το θέμα φυσικό ή πρόσωπο. Μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τον Επίτροπο να αναφερθεί στις ΕΠΟ, στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή, ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον έχει τονιστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κατάχρησης και διαφθοράς και απάτης. Το ανέφερε και συνάδελφος άλλωστε. Και έχετε δίκιο για αυτά που είπατε για τον, την Όλαφ. Επίσης, ό,τι αφορά τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, σίγουρα θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, ξανα συμβούν αυτά που όλοι έχουμε ακούσει. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Έχουν δοθεί περίπου, περίπου 5 ή και περισσότερα δισεκατομμύρια ευρώ σε μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, και δεν υπάρχει διαφάνεια σχετικά με την ε, χρήση τους. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μια διαδικασία στο ψηφιακή για να δούμε τι γίνεται με τα χρήματα που πηγαίνουν σε μη κυβερνητικέ οργανώσει, σε τρίτες χώρες για διάφορου ε, λόγους μέσω αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Χρειάζεται λοιπόν αύξηση της διαφάνειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ δεν πρόκειται για θέμα καχυποψία. όλοι θέλουμε να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα λεφτά μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους Ζεντόσκι, Κρότας και Γκραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε με πρόεδρε, ξέρετε με σκιώδεις εισηγητές. Πάρα πολύ προσεκτικά άκουσα τις παρατηρήσεις σας σε σχέση με την έκθεση αυτή και νομίζω ότι ε, μπορώ να είμαι ικανοποιημένο από τις αντρές γραμμές αυτής της έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ιδίω τα κεφάλαια που αφιερώνται στα διάφορα εξειδικευμένα ζητήματα. Σίγουρα ε, μπορούμε να βελτιώσουμε και κάποια σημεία με τροπολογίες. Αναφέρθηκαν και άλλοι ε, συνάδελφοι σε κάποιες τα οποία θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή ή λιγότερη έμφαση. Αλλά νομίζω αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε παντού ε, το ίδιο πρότυπο, το ίδιο κανόνα μέτρηση. Θα ευχαριστήσω και τον ε, Επίτροπο Χάν γιατί μίλησε με μεγάλη ειλικρίνεια και ανοιχτό πνεύμα τα προηγούμενα πέντε χρόνια δεν είδα ε, η Κομισιόν ε, να αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα. Η συγγήτρια ανέφερε συγκεκριμένα σημαντικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη θέλουμε ένα ψηφιακό μητρό για τους δικαιούχους ε, των επιδοτήσεων. Όχι σε ό,τι αφορά το που κάποιος μπορεί να έχει την επίσημη εγκατάσταση έντρα του, αλλά πραγματικά να βλέπουμε ποιος παίρνει τα χρήματα. Αυτό πρέπει να αναζητήσουμε. Ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος. Και σίγουρα δεν θα πρέπει στο τέλος της όλης αλυσίδας να βρίσκεται ένας ολιγάρχης ή με ολιγαρχική ομάδα ή δομή θα συμφωνήσω και με τον Ολιβιέ Σαστέλ που λέει ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και θα πρέπει να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Πρέπει να κατονομάζουμε, Ολιβιέ, όμως εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου γιατί έτσι ε, μπορούμε να ε, αποτρέψουμε ε, την επανάληψη. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιοριστούμε σε γενικολογίες θα πρέπει να μην περιοριζόμαστε σε γενικόλογες συστάσεις, αλλά να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και μας τα λέει και το ελεγκτικό συνέδριο, μας λέει τα ποσοστά ασφάλματος 5, 3,5, 3,7 και του λέμε μπράβο που τα εντόπισε το ελεγκτικό. Όχι, δεν αρκεί αυτό, είμαστε πολιτικοί και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα, να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και κάτι άλλο στο οποίο πιστεύω πρέπει να εστιάσουμε είναι τι γίνεται με τα κονδύλια τα οποία εκταμιεύονται από το μικρό μας ε, προϋπολογισμό. Να δούμε τι προστιθέμενη αξία έχουν, αν έχουν. Έχουν προστιθέμενη αξία στα κρατη Και τελικά να μην βοηθήσει ε, η χρηματοδότηση κάποιους συγκεκριμένους ε, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, δεν ξέρω που να πολλαπλασιάσουν, να αυγατήσουν τα λεφτά τους. Θέλουμε καλύτερο έλεγχο, καλύτερο έλεγχο για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εξού και κάνουμε ε, όλες αυτές τις κάνουμε όλου αυτού του ελέγχου και έχουμε τη διαδικασία χορήγηση απαλλαγή. Βλέπουμε τι γίνεται και στου εκτελεστικού οργανισμού. Θέλουμε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Θέλουμε να μην υπάρχει απάτη, διαφθορά. Γι' αυτό θέλουμε συγκεκριμένου κανόνε. Μόνο έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Βόλτε, επόμενο στο κατάλογο. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ με τη σειρά μου ένα ζήτημα. Ο Επίτροπος μα είπε ότι πρέπει να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Πολύ ωραία, συμφωνώ με αυτό. Και το αναφέρετε κι εσεί, Πρόεδρε, στην εκθεσή σα το ζήτημα αυτό. Αναλύεται εκτενώς το ζήτημα τη σύγκρουση συμφερόντων. Και λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταπολεμήσει κάθε μορφή σύγκρουση συμφερόντων. Και αναφερθήκατε κι εσεί, κυρία Πρόεδρε, σε ένα σχετικό άρθρο των New York Times νομίζω ότι σαφώς θα πρέπει να γίνεται μία αναφορά στο ζήτημα αυτό και στη δική σας την έκθεση. Ωστόσο, το άρθρο του New York Times αναφέρεται σε κάποιες τροπολογίες ε, της Επιτροπής Άγκρη, οι, οποία όμως, οι οποίες όμως ε, καταψηφίστηκαν από το σώμα της ε, Ολομέλειας. η τροπολογία αυτή αναφέρεται σε σύγκρουση συμφερόντων όχι μόνο από την εθνική σκοπιά, αλλά όταν αυτή προκύπτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε ότι πολύ συχνά στα πλαίσια της τροπολογίας αυτής γίνεται αναφορά στα φαινόμενα αυτά που έχουμε για σύγκρουση συμφερόντων, ακόμη και φαινόμενα διαφθοράς, από δημόσιους λειτουργούς σε εθνικό, περιφερειακό ή ακόμη και τοπικό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Προφανώς δεν θα πρέπει να έχουμε δικαιούχους στο πλαίσιο των γεωργικών ταμείων οι οποίοι έχουν περάσει από τέτοια καθεστώτα διαφθοράς. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμείνουμε στο ζήτημα αυτό των πολιτικών εκείνων που έχουν καταρτήσει συγκεκριμένου κανόνες και που έπειτα δεν τους στηρούν ή πολιτικοί οι οποίοι έχουν καταρτήσει κανόνες και είναι παράλληλα και οι δικαιούχοι συγκεκριμένων κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί προφανώ έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει εκ νέου να αναλύσουμε το ζήτημα αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή τη στιγμή μια ανοιχτή συζήτηση. Θέλουμε και εμεί να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Πάντω υπάρχει μια σχετική τροπολογία από την Επιτροπή Γεωργία. Θα πρέπει και αυτό να το έχετε υπόψη, κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκραπίνη. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξ αρχής ε, πρέπει να πω ότι είναι πολύ θετική η έκθεσή σας. Δεν είναι μία απλή έκθεση απαλλαγής, είναι μία πλήρης σφαιρική έκθεση, κυρία Πρόεδρε. Και ως εισηγήτρια πραγματικά αναφερθήκατε σε πολλά διαφορετικά και σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν όμως και στο μέλλον. Βασικό στόχος άλλωστε μιας απαλλαγής είναι να γίνεται η κατάλληλη ανάλυση και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές που ανέφερε και ο Επίτροπος. Γνωρίζω τον Επίτροπο ήδη από το 2012 όταν ήμουν υπουργό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μου και πραγματικά του έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Αναφερθήκατε στα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αναφερθήκατε σε πανεπιστήμια, σε αυτή την πλευρά της Ευρώπης, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με την καινοτομία και δεν τη χρησιμοποιούν ακόμα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την ε, έρευνα αυτή που γίνεται από τα πανεπιστήμια με την έρευνα που γίνεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δεν το έχουμε επιτύχει ακόμα και πολλές φορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι καινοτόμες, βρίσκονται κάπως περιθωριοποιημένες και απομονωμένες. Είναι πραγματικά θλιβερό νομίζω να επιτελείται ένα τόσο σημαντικό έργο έρευνα από τα πανεπιστήμια και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και έπειτα αυτό να μην αξιοποιείται. Ενδεχομένω στο μέλλον κυρία Πρόεδρε, ακόμα και στη δική σα την έκθεση, να μπορείτε να αναφέρετε λίγο περισσότερο τη σημαντικότατη αυτή διασύνδεση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ερευνητικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σαφώ θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την έρευνα η οποία επιτελείται, όπω σα είπα, και από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μία ακόμα πτυχή που θίγεται, κυρία Πρόεδρε, και αυτό με ικανοποιεί όλου ιδιαιτέρω, είναι ότι αναφέρεστε στον μηχανισμό αυτό που θα πρέπει να ισχύει για τους αγρότες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σύστημα υποβολής καταγγελιών από τους μικρούς ή μικρομεσαίους αν θέλετε αγρότες. Οι περισσότεροι εκ των οποίων φοβούνται να υποβάλουν καταγγελίες γιατί φοβούνται πως καταλήξουν τελικά σε ένα μαύρο κατάλογο. Νομίζω ότι θα πρέπει να τους ενισχύσουμε και να τους πλαισιώσουμε και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση το έθιξε εν μέρη και ο Επίτροπο αναφερόμενος σε αυτό το corporate register, το εταιρικό μητρό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει. Όσον αφορά τώρα τους τελωνιακούς δασμούς, έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία υπερασπίζεται τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα μπορεί να, αποτελέσει, να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω όμως ότι ε, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οργανισμοί μέσω του έργου τους να καταφέρουν τελικά να μειώσουν τα επίπεδα διαφθοράς και απάτης που έχουμε για την συλλογή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αν καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ τον κοινοτικό προπολογισμό. Κάτι τελευταίο το οποίο θέλω να θίξω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο Επίτροπος σε σχέση με την συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει κάθε φορά να έχουμε τι σωστέ πληροφορίε, τα σωστά δεδομένα, αν δεν καταφέρνουμε να συλλέγουμε και να αντλούμε τα κατάλληλα αξιόπιστα δεδομένα από τα κράτη-μέλη, τότε το τελικό αποτέλεσμα προφανώ δεν θα είναι θετικό όσον αφορά την αποτίμηση του ε, προπολογισμού. Ορισμένοι ρίχνουν μόνο την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το ένα, δήλωσε το άλλο και το καθεξής. Αυτό πολλέ φορέ όμω δεν είναι αντικειμενικό. Πολλέ φορέ λαμβάνουμε και εμεί λανθασμένες αποφάσεις μόνο και μόνο επειδή βασιζόμαστε σε εσφαλμένες πληροφορίε. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον Επίτροπό μα και στη δική μα την Επιτροπή. Ξέρετε ότι η έκθεση αυτή σίγουρα θα συμβάλλει σε μια βελτίωση τη υφιστάμενη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκραπίνη. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει ένα μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό ε, και βοηθά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ε, χρησιμοποιήσουν τα ερευνητικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια είναι κάτι για το οποίο παλεύει συνέχεια η Επιτροπή Προϋπολογισμών να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα κονδύλια. Κυρία Βόλτερς, όταν ε, τίθεται θέμα ψηφοφορίας ε, για τους ε, ευρωβουλευτές νομίζω πως χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή γιατί υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι που είναι του επαγγέλματο, προέρχονται από τον χώρο της γεωργίας και υπάρχουν πραγματικά συστημικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την όλη διαδικασία. Όταν ε, κάποιος είναι αγρότης και έχει 100 εκτάρια και λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις, αυτό καθιστά ε, θέμα επιρροής ή όχι. Είναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα και χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουμε. υπάρχουν ορισμένοι τομείς οι οποίοι δεν είναι μόνο πολιτικά ευαίσθητοι αλλά και ουσιαστικά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθούν τρόποι να αυξηθεί η διαφάνεια, η ψηφιοποίηση όπως είπε ο συνάδελφος Αστέλη είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα διευκολύνει την πρόσβαση σε όλους. Χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων από και στην ε, κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και φυσικά υπάρχει ανάγκη για ένα εναρμονισμένο σύστημα που θα χρησιμοποιούν όλοι, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα. Θα χρειαστεί λοιπόν να γίνουν αρκετές συζητήσεις έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την ε, Κομισιόν στην προσπάθεια αυτή. Αλλά να ξέρουμε γιατί μιλάμε, για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Οπότε λοιπόν ε, τονίζω πως ε, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές και τους βοηθούς τους, όλες τις πολιτικές ομάδες που βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά και την γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, την Αν ε, Κατρίνη η οποία βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση για το σημείο 3 και περνάμε στο σημείο 4 στην απαλλαγή Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Χάν που ήρθε και θα δώσω τον λόγο στην κυρία Γκραπίνη αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Στην πρώτη μας λοιπόν αυτή συζήτηση και καθότι είναι και η πρώτη συνεδρίαση μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους ένα πολύ ευτυχισμένο νέο έτος. Στην έκθεσή μου αυτή προσπάθησα να λάβω υπόψη μου και τις πραγματικές απαιτήσεις και προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Καταρχάς όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία η οποία με υποστήριξε όλους ιδιαίτερως κατά την κατάρτιση της έκθεσής μου αυτής. Ως βασική συγκήτρια για το ζήτημα αυτό κατάφερα μέχρι τα τέλη του 2019 να ολοκληρώσω το σχέδιο του κειμένου όσον αφορά την απαλλαγή για το έτος 2018 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο του σχεδίου έκθεσης κάναμε κάποιες ακροάσεις με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βέλε, του κ. Σίλβα Περέιρα και είχαμε επίσης και τη βοήθεια των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου και ως εισηγήτρια συνάντησα εκπροσώπους από 12 γενικές διευθύνσεις. Πέρασα λοιπόν πάρα πολύ χρόνο και κατέβαλα αρκετές προσπάθειες για να καταφέρω να καταρτήσω την έκθεση αυτή που έχετε ενώπιον σα και βέβαια συναντήθηκα και με του εκπροσώπου του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ θετική η εμπειρία που είχα όταν χρειάστηκε να εντοπίσω κάποια προβλήματα τα οποία είχε αναφέρει ο Γενικό Γραμματέα, αλλά και το προσωπικό του Κοινοβουλίου και με ιδιαίτερη χαρά είδα ότι είχε σημειωθεί μια κάποια βελτίωση και μια κάποια πρόοδο. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλε τι γενικέ διευθύνσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίε ήταν ιδιαίτερα διαλλακτικέ και μίλησαν ανοιχτά μαζί μου. Καταλήγω εδώ σε κάποια συμπεράσματα και σε κάποιες συστάσεις βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο και καταλήγω και σε κάποια δικά μου συμπεράσματα που αποτελούν ε, αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαμε εκπροσώπους του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θίγονται πολλά ζητήματα στην έκθεση αυτή που έχουν να κάνουν με τις επιμέρους γενικές διευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν γέννη πάντως μπορούμε να πούμε ότι η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει βελτιωθεί, ιδίως προς το τέλος της προηγούμενης νομοθετικής εντολής. Χρειάστηκε, ιδίω το τελευταίο έτος, να ασχοληθούμε με πολλά διαφορετικά ζητήματα, με έναν αυξημένο φόρτο εργασία. Η απόφαση του Μένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει ποικιλοτρόπω ε, τι γενικέ διευθύνσει ε, του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχει επίσης και το, ο στόχος της μείωσης κατά 5% του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι χρειάστηκε να καταργηθούν 60 θέσεις απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια μέση διασύνδεση βέβαια ανάμεσα στο μεγάλο αριθμό ε, αδειών ανάρρωσης που έχουν δοθεί και στον ε, αριθμό μείωσης του προσωπικού οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνέχισαν τελικά να εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρέθηκαν επιφορτισμένοι με ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε σε ορισμένες άδειε ασθένειας. Επίσης, στα πλαίσια της έκθεσής μου τονίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή και ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξορροπήσουν προσωπική και επαγγελματική ζωή. Διότι καταλαβαίνετε ότι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τελικά οι γενικές διευθύνσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο τελικά επηρεάζει και το δικό μα το έργο, το έργο των Ευρωβουλευτών δηλαδή. Επίση, στην έκθεσή μου αναφέρομαι στι δραστηριότητε εκείνε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίε ε, είναι πολύ σημαντικέ για την ε, λειτουργία του δικού μα ε, του έργου, ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να προσλάβουμε προσωπικό από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο Γενικό Γραμματέα να καταβάλει προσπάθειε προκειμένου να υπάρχει η κατάλληλη γεωγραφική κατανομή όσον αφορά το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει το προσωπικό αυτό να εκπροσωπείται βέβαια ισότιμα και στις διευθυντικές θέσεις. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει βέβαια και για την ε, ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και σε διευθυντικές προφανώς σχέσεις. Θα πρέπει να μας απασχολεί η πτυχή αυτή της διάστασης του φύλου σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει μέσω συγκεκριμένων μέτρων να επιβάλλουμε τον δικό χάρτη για την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να έχουμε όλο και περισσότερες ε, γυναίκες διευθυντές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι τα τέλη του 2019 οι στόχοι μας στον τομέα αυτό δεν είχαν ακόμα επιτευχθεί και γι' αυτό το λόγο προτείνω ο στόχος αυτός να παραμείνει και για το 2020 αλλά και για τα επόμενα χρόνια μέχρι τελικά να επιτευχθεί αυτή η ισότιμη εκπροσώπηση σε διευθυντικέ θέσεις ανδρών και γυναικών. Επίση, ερχόμενοι σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, είδα ότι υπάρχουν ορισμένα κρατημέλη τα οποία δεν εκπροσωπούνται καθόλου σε επίπεδο διευθυντή ή γενικού διευθυντή και νομίζω ότι ε, και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επιληθεί. Όσον αφορά επίσης του διερμηνείς, Καταλαβαίνουμε τι συνέβη με τι συνθήκε εργασία του. Κάποια στιγμή όμω, την προηγούμενη μα εντολή, είδαμε ότι υπήρχε μία σύγκρουση ανάμεσα στου διερμηνεί και την ε, αρμόδια διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία η κατάσταση αυτή καθώς επίσης και η κατάσταση των μεταφραστών. Αυτοί υπεργάζονται δηλαδή στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, οι οποίοι βρέθηκαν υπό έναν υπερβολικό φόρτο εργασίας λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας στο τέλος της θητείας, αλλά και λόγω των νέων καθηκόντων που καλούνται να επιτελέσουν τώρα. Γι' αυτό το λόγο κάλεσα τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη από τη διεύθυνση αυτή να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να ασχοληθούμε λίγο και με το ζήτημα της ποιότητας προσωπικής ζωής των εργαζομένων αυτών. Επίσης, ε, ε, χρειάστηκαν οι διευθύνσεις αυτές να αντιμετωπίσουν ε, το φαινόμενο του περιορισμένου προσωπικού που έχουν. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται να τα φέρουν εις πέρας με περιορισμένο προπολογισμό. Και το θέμα είναι ότι οι περιορισμένοι προπολογισμοί πολλές φορές στις διάφορες γενικές διευθύνσεις προκαλούν πολλά προβλήματα και στους εργαζόμενους. Όσον αφορά την ε, αποζημίωση, καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Πρέπει να είναι κανεί πάρα πολύ αυστηρό όσον αφορά το ζήτημα των αποζημιώσεων και ε, είχαμε κάποια προβλήματα, ιδίω με το Γραφείο Ταξιδίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο Γραφείο Ταξιδίων που συνεργάζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Γίνανε κάποια παράπονα, κάποιε καταγγελίε. Γι' αυτό το λόγο στην έκθεσή μου προτείνω και κάποια μέτρα βελτίωση τη δραστηριότητα του γραφείου αυτού. Υπάρχουν διάφορε καθυστερήσει, όπω σα είπα, όσον αφορά την κάλυψη των ταξιδιωτικών δαπανών. Όσον αφορά τώρα την Γενική Διεύθυνση Καινοτομία και Τεχνολογική Υποστήριξη, τη Γενική Διεύθυνση ΙΤΕΚ, υπήρξαν εδώ προβλήματα στην πρόσληψη ειδικευμένου, υψηλά ειδικευμένου προσωπικού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να λάβει υπόψη το αίτημα της Γενικής αυτής Διεύθυνσης προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλε προσλήψεις. Θα πρέπει ουσιαστικά η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες και κενά όσον αφορά την λειτουργία του δικτύου ίντερνετ, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά της ψηφιακή υποδομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα και θα πρέπει η Γενική Διεύθυνση ETEC να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον ψηφιακό τομέα. Μάλιστα, πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Γενική αυτή Διεύθυνση προχώρησε σε μία ανακοίνωση που εστέφθη με επιτυχία και είδαμε ότι υπήρχε τελικά και μια πολύ έντονη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωπαϊκές εκλογές. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, της Γενικής Διεύθυνσης ΚΟΜ. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο τη στρατηγική επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, να είναι πιο προβεβλημένη και πιο προσβάσιμη από του Ευρωπαίου πολίτε. Τώρα, η συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ξέρετε ότι είναι μια ιδέα η οποία προέκυψε από το ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι αρκετά κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, Ξέρουμε ότι έχουμε τα γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα λεγόμενα e Θα πρέπει και αυτά να εμπλακούν περισσότερο προκειμένου να φέρουν πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ευρωπαίου πολίτε. Υποστηρίζω επίση τι προσπάθειε τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Λικοτεχνική Υποστήριξη τη Γενική Διεύθυνση ΙΝΛΟ, προκειμένου να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλεια. Πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί προ του πολίτε εγγυόμενοι όμως και την ασφάλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 142 είναι τα σημεία τα οποία παριθμεί η έκθεσή μου, δεν θα ήθελα να αφαιρθώ σε καθένα από αυτά. Εν κατακλείδη μόνο να σας πω ότι η όλη εμπειρία κατάρτισης έκθεσης αυτής ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τη γραμματεία. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να έχω όλες αυτές τις επαφές και τις συζητήσεις με τις Γενικές Διευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, προσβλέπω στις δικές σας παρατηρήσεις η, ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών 29 Ιανουαρίου. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μια θετική έκθεση η οποία θα βελτιώσει πραγματικά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκραπίνη. Ο Τάμας Ντόιτς έχει τώρα το λόγο ως και ο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, η έκθεση είναι φέτος ε, πιο λεπτομερής και στο όνομα του ΕΛΚ λοιπόν καλωσορίζω την έκθεση. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι γνωρίζουμε όλοι πώς μπορούμε να υποβάλουμε γραπτές ερωτήσεις αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα ικανοποιητικέ απαντήσεις από Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Ε, κατά την ε, συνεδρία της ομάδας ελέγχου του προϋπολογισμού ήταν παρόν, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Εμείς θεωρούμε πως οι απαντήσεις ήταν ικανοποιητικές. Καλωσορίζουμε και την κατεύθυνση της έκθεσης αυτής. παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ίσως ε, χρειαστούν ορισμένες τροποποιήσεις. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και να πω ότι θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Δεν θέλω να πω εδώ ότι πρόκειται για παράπονα από ορισμένους ευρωβουλευτές, αλλά υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν την χρήση των ε, κονδυλίων. Το ΕΛΚ, λοιπόν, θεωρεί απαράδεκτο ότι, για παράδειγμα, το ταξιδιωτικό πρακτορείο του Κοινοβουλίου που έχει σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ε, πιο ακριβά εισιτήρια από αυτά που μπορεί να βρει κάποιος ε, ψάχνοντας μόνος του. Μιλάμε για αεροπορικά εισιτήρια ή για εισιτήρια τρένου. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο και μικρό, όμως ε, μετά το Brexit θα έχουμε πάνω από 700 ευρωβουλευτές οι οποίοι δουλεύουν 40 εβδομάδες το χρόνο, πρέπει να ταξιδεύουν συνεχώς και στα Ουγγρικά έχουμε και μια παροιμία που λέει ότι και το μικρό βοηθά και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάνουμε κάτι έστω για να διορθώσουμε τα μικρά προβλήματα, νομίζω πως θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω με τις τροπολογίες μου να είμαι σαφής. Η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλο το ταξίδι από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο ή από τις ε, πατρίδες μας στο Στρασβούργο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί επιτέλους, να υπάρχουν σαφείς όροι. Είμαι εδώ από το 2009 και για πάρα πολλά χρόνια συζητιόταν το θέμα της ε, έδρας του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να φύγει το Κοινοβούλιο από το Στρασβούργο. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες και δεν το θεωρώ πολιτικά εφικτό στην παρούσα στιγμή. Το θέμα της ενιαίας έδρας του Κοινοβουλίου είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, όμως η κατάσταση πώς έχει. Είτε θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει το δικαίωμα να το κάνει, ότι θα φύγει από τις Βρυξέλλες και θα μετακομίσει εξ ολοκλήρου στο Στρασβούργο. Φυσικά και μπορεί να το αποφασίσει αυτό το κοινοβούλιο. Μιλάμε για κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ή στην περίπτωση που αποφασίσει το αντίθετο, να μετακομίσει εξ ολοκλήρου στις Βρυξέλλες και να σταματήσουμε το, να πηγαίνουμε στο Στρασβούργο. Είναι θέμα κόστου. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογιστεί το κόστος και στις δύο περιπτώσεις έτσι ώστε να ε, σταματήσουν πλέον αυτά τα πηγενέλα μεταξύ των δύο εδρών. Φυσικά υπάρχει επιχειρηματολογία και για τις δύο περιπτώσεις, όμως δεν νομίζω να καταλήξουμε σύντομα σε κάποια απόφαση. Αυτό το θέμα λοιπόν ε, με το πηγενέλε και τις δύο έδρες νομίζω πρέπει επιτέλους να μας απασχολήσει για να βρεθεί μια λύση. Νομίζω πως είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι θα λυθεί σύντομα. Και ωραία είναι να λέμε μακάρι να γινόταν κάτι, όμως αυτό δεν είναι πραγματικότητα προς το παρόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διερμηνία, η απάντηση του Γενικού Γραμματέα πώς να το πω, δεν ε, μας λύνει και τελείως ε, το πρόβλημα. Νομίζω πως ε, βρισκόμαστε ακόμα σε κάποια διαφωνία. Υπάρχει κόστος για τη διερμηνία που διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα. Για παράδειγμα, μία ώρα διερμηνία στα Ισπανικά κοστίζει 500 ευρώ, μία ώρα διερμηνία στα Ρουμάνικα 250 ευρώ. Εντάξει, είναι φυσιολογικό αυτό, διότι πιο πολύ μιλούν Ισπανικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρουμάνικα. Όμως, αυτό οδηγεί σε ορισμένες διαφορές. Για παράδειγμα, οι διερμηνείς της ισπανικής γλώσσας είναι ανήκουν σε υψηλότερη βαθμίδα από ό,τι διαμηνείς τη ρουμάνικης γλώσσας ή παρομοίως για τα μαλτέζικα και τα αγγλικά. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν οι οποίες δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμα σε ό,τι αφορά ε, το, την ε, διερμηνία. Έπειτα, η, η συγγήτρια αναφέρθηκε στις ε, γεωγραφικές διαφορές. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητάμε συχνά. Χωρίς όμως να πλησιάζουμε στη λύση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω το εξή. Το 2009 υπήρχαν 10 κράτη-μέλη παραπάνω. Τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Όμως το 2009 είχαμε μόνο δύο Πολωνούς οι οποίοι ήταν επικεφαλής τμήματων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ λίγοι. Στο μεταξύ οι δύο έχουν γίνει έξι το 2019 όμως υπάρχει ακόμα μία άνηση εκπροσώπηση. Υπάρχουν λιγότεροι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι από τις νέες χώρες. Τώρα, στους ε, διοικητικούς υπαλλήλους της βαθμίδας AD9 υπήρχαν 30 άτομα από τις νέες χώρες. Όχι, 30 άτομα γενικότερα. Από τα 30 άτομα, οι 10 ήταν Γερμανοί και οι 6 ήταν Ιταλοί. Οι υπάλληλοι λοιπόν από τις νέε χώρες ήταν λιγότεροι από τους Γερμανούς υπαλλήλου. Πρέπει λοιπόν η κατάσταση να αλλάξει. Το 2014 προσθέθηκαν ακόμα περισσότεροι Γερμανοί, ακόμα περισσότεροι Ιταλοί και η εκπροσώπηση από Ούγγρους, ας πούμε, Μαλτέζους, Κύπριους ήταν πάρα πολύ ε, χαμηλή και η δικαιολογία ήταν ότι δεν είχαν τα προσόντα ε, για να στελεχώσουν τις θέσεις αυτές, αυτού του βαθμού. Τώρα θα ήθελα κλείνοντα να ευχαριστήσω ξανά την εισηγήτρια και ε, να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Τσιλμπογιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία. Πραγματικά χρειάστηκε να καταπονήσετε πάρα πολύ εργασία προκειμένου να έχουμε μια τόσο πλήρη και σφαιρική έκθεση. Η δική μου πολιτική ομάδα μέσω του υποφαινούμενου θα καταβάλει, καταθέσει κάποιες τροπολογίες, θα ήθελα να εστιαστώ σε τρία σημεία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά πρώτον. Είναι πολύ σημαντικό και το θίξαμε αυτό και στην προηγούμενη συζήτηση ότι θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια των θεσμικών μας οργάνων. Αυτό είναι μια δημοκρατική απέτηση το θίξαμε πάρα πολύ ορισμένοι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκλογικής εκστρατείας και κατά αυτόν τον τρόπο θα συμφιλιώσουμε τρόπον την τον Ευρωπαίο πολίτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμικά της όργανα. Και δύο εκθέσεις στις οποίες αναφερθήκατε δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ αλλά αποτέλεσαν μόνο αντικείμενο διαβούλευσης και κλεισμένων των θυρών ανάμεσα σε ευρωβουλευτές. Καταλαβαίνετε όμως ότι κάθε φορά που συνεδριάζουμε με απόρριτες εκθέσεις και κλεισμένων των θυρών, πολύ συχνά συνειδητοποιούμε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος οι συνεδριάσεις αυτές να είναι τόσο μυστικές και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μία αδικαιολόγητη περιττή καχυποψία στους Ευρωπαίους πολίτες, ανεφλόγου και αιτίας. Και να σκέφτομαι για παράδειγμα την, την έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή θα μπορούσε να αναφερθεί κανείς και στην έκθεση του αρμοδίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Για ποιο λόγο οι εκθέσεις αυτές να μην είναι δημόσιες. Κάτι το οποίο θίξατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε στην εκθεσή σας, στην παράγραφο 31 συγκεκριμένα, όσον αφορά την κατάργηση θέσεων απασχόλησης στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάργηση θέσεων απασχόλησης δεν είναι προφανώς ποτέ ένα θετικό νέο και σε ορισμένες περιπτώσεις διερωτάται κανείς για τον φόρτο εργασία που απομένει για αυτούς οι οποίοι θα παραμείνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αναφέρετε και εσείς αυτό λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μερικές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την κατάργηση θέσεων απασχόλησης λέγοντας ότι αυτό γίνεται για λόγους εξορθολογισμού ή εξοικονόμησης, ιδίως όταν αναφερόμαστε στα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Σαφώς πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση όμως των θέσεων προς κατάργηση, να γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο καταργούνται και πώς η συνέχεια μπορεί να εξορροπηθεί ο αναπαμείνων φόρτος εργασίας. Γιατί το να παρουσιάζουμε απλώς το ζήτημα αυτό ως μια ανισχυτική εξέλιξη, σαφώς μπορεί να μας ανισχύει το φαινόμενο αυτό, αλλά ενδεχομένως να είναι και δικαιολογημένε τελικά οι καταργήσεις κάποιων θέσεων απασχόλησης. Και ένα ακόμα σημείο, το οποίο δεν μπορώ παρά να το θίξω, το ζήτημα της διπλής έδρας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο κύριος Ντόιτς πριν από λίγο το έθεσε το ζήτημα αυτό. Ξέρετε ότι κάθε άρθρο της συνθήκης αντιστοιχεί και σε ένα κόστος, όχι μόνο το συγκεκριμένο αυτό άρθρο. Θα σας πρότεινα λοιπόν αν θέλετε να αποτιμήσουμε το κόστος όλων των άρθρων της συνθήκης και όχι μόνο αυτού του συγκεκριμένου άρθρου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να απομονώνουμε μόνο αυτό το άρθρο και να λέμε η συγκεκριμένη δέσμευση συνθήκη μας στοιχίζει τόσα ευρώ, ενώ μπορεί να υπάρχουν άλλα άρθρα τα οποία να αντιστοιχούν σε πολύ υψηλότερο κόστος. Ενδεχομένω σα προκαλώ αυτή τη στιγμή και σα ζητώ συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να πω και το ακόλουθο. Εφόσον η έδρα του Κοινοβουλίου βρίσκεται στο Στρασβούργο, μήπω θα έπρεπε να αποτιμήσουμε πόσο στοιχίζει τον να ερχόμαστε στι Βρυξέλλε, γιατί η επίσημη έδρα του Κοινοβουλίου είναι στο Στρασβούργο. Α μην το ξεχνάμε αυτό. Σα προκαλώ και μια δεύτερη φορά τώρα και ενδεχομένω να στοιχίζει πολύ περισσότερο να ερχόμαστε στι Βρυξέλλε από ότι να πηγαίνουμε στο Στρασβούργο. Τούτων λεχθέντων, ξέρω το ζήτημα είναι πολύ ευαίσθητο, ξέρω ποια είναι η θέση των υπόλοιπων συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια είναι η θέση τη γαλλική αντιπροσωπεία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το να απομονώνουμε το άρθρο αυτό της συνθήκης, να εστιαζόμαστε μόνο στο άρθρο αυτό και να αποτιμούμε το κόστος των αποστολών προς το Στρασβούργο, ενώ το Στρασβούργο είναι η επίσημη έδρα του Κοινοβουλίου, για μας είναι κάπως προκλητικό, πώ να το πω διαφορετικά. Και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σχετική μνήα στην έκθεση αυτή. Ξέρω ότι βρίσκομαι στη μειονότητα λέγοντα κάτι τέτοιο. Παρ' αυτά έπρεπε να το θίξω και θα υποβάλω και σχετικέ τροπολογίε. Σα ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν να προχωρήσουμε με τους άλλους ε, συνάδελφους που έχουν στήσει το λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι η Σύμβαση της Λισαβόνας ε, τα λέει κάθαρα με το πρωτόκολλο 8 για τι συνθήκε πρωτοξιανουσία. Με έχει απασχολήσει αυτό το θέμα αυτό και θα μπορούσα να το επαναλάβω ότι εκεί γίνεται λόγο για τρει ε, τόπου εργασία και αναφέρονται όλοι οι τόποι εργασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινομούλιο μπορεί να πάρει ακόμα 5.000 φορές την απόφαση να πάει αλλού την έδρα του, αλλά χρειάζεται ομοφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου για να αλλάξει το τίποτα. Μπορούμε 500.000 φορές να τα συζητήσουμε και να τα ε, κατηγορούμε και να τα καταγγέλουμε όλα αυτά, αλλά... Ε, ε, τι να πούμε, η μισή λένε Βρυξέλλες, η άλλη μισή Στρασβούργο και τα δύο είναι πολύ ωραία αλλά δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει ούτε την Επιτροπή μας ε, αυτό. Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι αυτός ο υπολογισμός ε, του κόστους που λέτε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υπερφορτώσουμε τη διοίκηση με στη δουλειά. Ε, δηλαδή ε, τι θα κόστιζε αν κάποιος πετάει για Βρυξέλλες ή αν κάποιος πετάει για Στρασβούργο. Για μένα θα ήταν πιο φτηνό το Στρασβούργο ε, που είμαι κοντά. Για άλλους είναι πιο μακριά. Δηλαδή μην μπαίνουμε σε τέτοιες ασκήσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα και λογική. Και θα δώσω το λόγο, δεν ξέρω αν ο συνάδελφος Πέξα στη θέση του συνάδελφου Φρόντ θα πάρει συνέχεια το λόγο, αλλά να προσθέσω και κάτι τελευταίο, ότι ε, υπάρχει ένα θέμα με τα αυτοκίνητα τα οποία ε, ταξιδεύουν, ε, οι λιμουζίνες αυτές, τα θα μπορούσαν πράγματι να παίρνουν και οι υπαλλήλου να φεύγουν πιο γεμάτα δηλαδή, γιατί μετά γεμίζουν τα λεωφορεία και βέβαια μένει ο κόσμος πολλή ώρα μέσα στο λεωφορείο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μπορούμε να το συζητήσουμε με το Προεδρείο για να είναι πιο αποδοτική η χρήση αυτών των υπηρεσιακών ε, οχημάτων. Αλλά ε, μην ε, δίνουμε έτσι εικόνες, έτσι, μην παρουσιάσουμε μια αρνητική βιτρίνα για το Κοινοβούλιο. Παναλαμβάνω. μπορούμε να το συζητήσουμε 500.000 φορές το θέμα της έδρας, αλλά αν δεν το αποφασίζει το Συμβούλιο, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε άλλες 500 φορές. Ε, πραγματικά ε, είναι λίγο κουραστικό να αποφασίζουμε εμεί συνέχεια ότι θέλουμε μία έδρα χ και να αποφασίζει τη έδρα και να πηγαίνουμε πέρα δόθε με το ε, αυτοκίνητο ή με τα μέσα για να ταξιδεύουμε. Λοιπόν, ας μην το ε, ξαναθέξουμε, να μην το ανοίγουμε αυτό το θέμα, ας εστιάσουμε στα θέματα που είναι δικής μας αρμοδιότητας. Εσύ, ο συνάδελφος Πέξα, που θα αντικαταστήσει αφοφρόιντ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστώ την κυρία Γκραπίνη για την έκθεση. Ο κύριος Φρόντινος και ο συγκητής δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Θα παρουσιάσω εγώ λοιπόν τη δική του άποψη. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του σχεδίου έκθεσης, ε, όπως παρουσιάστηκαν σήμερα, συμφωνούν με τη δική μας ανάλυση και εκτίμηση. Θα θέλαμε βέβαια από την ομάδα μας μεγαλύτερη ε, έμφαση σε κάποια σημεία που θεωρούμε ότι χρήζουν ιδιαίτερη πρόσοχη συγκεκριμένα. Η άποψη των Πρασίνων είναι πω ε, το ίδιο το Κοινοβούλιο είναι αυτό που θα πρέπει να παρακολουθεί πιο συστηματικά και το προτέρων του κανόνε περί διαφάνεια ηθική ε, και να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα στην ε, διαδικασία της ειδήσιας απαλλαγής. Επίσης, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να στηρίξει ε, τους βουλευτές, να τους δίνει φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα και εξοπλισμό πληροφορικής το lobby tool επίση είναι κάτι πολύ σημαντικό για να υπάρχει σχέση με το παρατηρητήριο και το μητρό διαφάνεια και, θα μπορούν να είναι μηχανοργανωμένο το περιεχόμενο. Επίσης, ε, ε, συμφωνώ ότι πρέπει να εστιάσουμε ε, στο να έχουμε μια ενιαία έδρα. Είναι προβληματικό το να ταξιδεύουμε κάθε μήνα. Είναι πολύ κουραστικό επίσης και χιλιάδες από εμάς να ταξιδεύουμε κάθε μήνα. Είναι περιβαλλοντικά παράλογο δε το να έχουμε έδρα σε δύο χώρες. Στην τελευταία έκθεση ε, δεν ε, έκανε το Προεδρείο τα δέοντα ε, σε σχέση με την αποζημίωση γενικών εξόδων. Ο Ντάινερ Φρόιντ αυτά θέλει να πει, αλλά εγώ θέλω να προσθέσω κάτι προσωπικά τώρα, από το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αλλάξει τον πάροχο υπηρεσιών στον Βρεφονδιακό Σταθμό το Φεβρουάριο. 3 Φεβρουαρίου είναι η αλλαγή αυτή. Και ανησυχεί το προσωπικό που απασχολείται αυτή τη στιγμή στον βρεφομιλιακό σταθμό, ανησυχεί και εμά που έχουμε τα παιδιά μα κάθε μέρα στο σταθμό αυτό. Επίση, αλλάζουν οι συνθήκες εργασίες, ε, το πρόγραμμα και μπαίνουν και άλλες αλλαγές εμείς θέλουμε το Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει ε, του και να αναφέρει στην αρμόδια επί της απαλλαγής ε, αρχή η ποιότητα ε, των υπηρεσιών για τα παιδιά μας ε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιδεινωθεί. Πρέπει να είναι φιλοκογενειακό το Κοινοβούλιο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος ε, από το ID το λόγο ή από την ομάδα ECR. Από την ΚΟΕ. Όχι. Πολύ ωραία. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει το λόγο η κυρία Γκραπίνη ξανά. Θέλετε να ακούσετε κάποιον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Η ε, Καταλήνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ σημαντικό το έργο όλων και των κοινοβουλευτικών βοηθών και τη γραμματεία και όλων. Θα, ήθελα να επαναλάβω ε, αυτό που είπε η Πρόεδρος, ότι το να σημειωθεί πρόοδος ε, σχετικά με τα ταξίδια κάθε μήνα στο Στραμβούργο είναι πολύ σημαντικό. Τα λεωφορεία που μεταφέρουν κόσμο πρέπει ε, να αρχίσουν να μεταφέρουν περισσότερους, πρέπει να μοιραζόμαστε το ταξίδι με το αυτοκίνητο και επίσης ε, θα χρειαστεί περισσότερη διαφάνεια στις αποζημιώσεις γενικών εξόδων. Συμφωνώ. Να υπογραμμίσω δύο σημεία. Από τη μία είναι πολύ θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, επιτευχθεί ουδετερότητα σε σχέση με τη χρήση άνθρακα μέχρι ε, το 2030. Ελπίζω λοιπόν να το δούμε και στο κείμενο αυτό. Θα καταθέσω και τις ε, σχετικές τροπολογίες ε, για το διοξίδιο του άνθρακα και επίσης ε, έχω να πω κάτι σχετικά με την εκπροσώπηση. Το κοινοβούλιο χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, βλέπω πολλούς νέους ευρωβουλευτές, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο. από τη στιγμή που εκλέγεται κάποιος ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παρνηθεί το δικαίωμά του να έχει παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ορίσει κάποιος ε, ο οποίος έχει γονική άδεια αντιπρόσωπο στις ε, ψηφοφορίες θα πρέπει να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ε, στις ε, ψηφοφορίες, το οποίο σημαίνει ότι όταν ε, κάποιος βρίσκεται σε γονική άδεια δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να ορίσει κάποιον στη θέση του. Αυτό νομίζω πως είναι κακό μήνυμα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που εκλέγονται σε αυτό το αξίωμα. Νομίζω λοιπόν πως έχει έρθει η ώρα να δείξει το Κοινοβούλιο πόσο προοδευτικό είναι και να αλλάξει αυτήν, ε, την, αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, ε, οι οποίοι νομίζω ότι εξέφρασαν πολύ ενδιαφέρουσες ε, ιδέες. Όπως σας είπα, τα 142 αυτά σημεία που βλέπετε στην εκθεσή μου αποτελούν απλώς σημεία ενός σχεδίου έκθεσης, το οποίο πρόκειται να βελτιωθεί βέβαια με τις δικές σας τις τροπολογίες, καθότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρω να συλλέξω πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό της απόκλησης Αποζημίωση τη απόκληση του κόστου τη διερμηνία από την μία γλώσσα στην άλλη. Ξέρετε ότι έχουμε ζητήσει επίσημα να υπάρχει το ίδιο επίπεδο αποζημίωση. Καταλαβαίνετε όμω ότι τα χρήματα τελικά τα οποία δίδονται στην διερμηνία έχουν να κάνουν με τι συνθήκε που ισχύουν στην αγορά διερμηνία, στην ιδιωτική αγορά διερμηνία κατά την πρόσληψη των freelance διερμηνέων. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται από τη μία καμπίνα στην άλλη ή από τον έναν γλωσσικό συνδυασμό στον άλλον. Και από ό,τι φαίνεται μερικές φορές το θεσμικό μας όργανο δεν είναι αρκετά ελκυστικό, διότι υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι επαγγελματίε οι οποίοι έχουν πολύ πιο υψηλές αποδοχές εργαζόμενοι στην ιδιωτική αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να καταστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ελκυστικό ως εργοδότη. Ενδεχομένως η ιδέα αυτή να περνούσε και σε μια τροπολογία. Θα ήταν καλή ιδέα αυτό. Η ε, απόκληση αυτή στις αποδοχέ έχει να κάνει όχι μόνο με τους διερμηνείς, αλλά και με τους βοηθού, τους τοπικούς μάλλον βοηθού των Ευρωβουλευτών. Θα πρέπει η τοπική βοηθή αλλά και η βοηθή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χαίρουν των ίδιων αποδοχών. Έπειτα, όσον αφορά τα πούλμαν, τα λεωφορεία, το είχαμε θίξει αυτό και με το Γενικό Γραμματέα. Για ποιο λόγο τα οχήματα αυτά να μην μπορούν να πάρουν και κάποιο από το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσαν τα οχήματα αυτά, ιδίως όταν πρόκειται για λεωφορεία, μικρά λεωφορεία, πέρα από τους ευρωβουλευτές να μπορούν να φιλοξενήσουν κατά το ταξίδι αυτό και άλλα μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά αυτόν τον τρόπο το ταξίδι γίνεται πολύ πιο αποδοτικό και λιγότερο ζημιογόνο για το περιβάλλον. Όσον αφορά το ζήτημα τη διαφάνεια, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια μυστικότητα όσον αφορά τι εκθέσει ελέγχου. Περιμένω απαντήσει και θα τι συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Να θίξω μία ακόμα πτυχή του ζητήματος. Το ανέφερε ο συνάδελφος από την ομάδα Renew Ως προς αυτό να πω ότι υπάρχει ένα κατόφλι κάτω από το οποίο δεν μπορεί να κατέβει κανείς αν θέλει να παραμείνει αποτελεσματικός. Αν μειώσετε τον αριθμό των εργαζομένων κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, πάβετε πλέον να είστε αποτελεσματικοί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην εξαφάνιση κάποιων θέσεων απασχόληση, αναφέρομαι στι επιπτώσει που εμεί οι ευρωβουλευτέ άμεσα θα αισθανθούμε. Ξέρετε ότι μερικές φορές προκύπτουν προβλήματα με το Wi-Fi, με τον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή εδώ πέρα στο γραφείο μου και χρειάζεται να περιμένω πάρα πολύ μέχρι να έρθει κάποιος τελικά να το επισκευάσει. Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, αλλά θα πρέπει να καταφέρνουμε να διατηρήσουμε και ένα χι επίπεδο εργαζομένων, προκειμένου να μπορούμε να εργαζόμαστε και αποτελεσματικά όσον αφορά τον βρεφονιπιακό σταθμό κάναμε μια σχετική συζήτηση με το Γενικό Γραμματέα και με τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Όντως υπάρχουν ορισμένοι ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν παραπονεθεί ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους στον βρεφονιπιακό σταθμό χρησιμοποιώντας α, τα μέσα τα οποία τους διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα είναι να δούμε τελικά αν μπορούμε να διατηρήσουμε την υπηρεσία αυτή. Ξέρετε ότι η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα δημογραφικό. Νομίζω ότι εμείς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτουμε περισσότερα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά. Θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν λοιπόν οι ευρωβουλευτέ ε, τα οχήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να πάνε τα παιδιά τους και στο βρεφονιπιακό σταθμό. Σε όλα τα ζητήματα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε και σε κάποιους συμβιβασμούς. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή απαλλαγής μπορεί πραγματικά να οδηγήσει μια βελτίωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσβλέπω λοιπόν στις δικές σας ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. όταν ε, λείπει ένας ευρωβουλευτής για τους οποιοδήποτε λόγους, επειδή έχει γονική άδεια, είτε επειδή είναι άρρωστος, δεν υπάρχει ε, και δεν προβλέπεται αντικατάστασή του από κάποιον άλλο. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Ε, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ και την εισηγήτρια, την κυρία Γκραπίνη, όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης και στην κυρία Ριβαζή. Πρόκειται για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω για την έκθεση ΕΤΑ, για το ΦΕΔ. Όπως προβλέπει η διαδικασία, βασίστηκα στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για επίσης τις ε, ερωταπαντήσεις ΔΕΦΚΟ και 28 Νοεμβρίου στην ανταλλαγή με τον Επίτροπο ε, Μίμητσα και στη γραπτή επίσης διαδικασία που ε, ακολούθησε με τον Επίτροπο Μίμητσα. Η Επιτροπή σήμερα θα γνωμοδοτήσει και θα γίνει και ψηφοφορία ποιες είναι οι ατρέ γραμμές της έκθεσης που είμαι βέβαιο ότι το ξεκοκαλίσατε το κείμενο, το έχετε διαβάσει αναλυτικά. Λέμε ότι πρέπει οι πολιτικές οι αναπτυξίε συνεργασίες να ευθυγραμμιστούν με τις αναπτυξιέ προτεραιότητε των χωρών εταίρων, δραστηριότητε του ΕΤΑ είναι μέσα σε ένα δύσκολο πλαίσιο και υπάρχουν γεωποκυλητικοί θεσμικοί επαναλαμβανόμενοι κίνδυνοι. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί τρόποι εφαρμογή, ένα ευρυφάσμα που δείχνει τη διακυβερνητική δομή του ΕΤΑ. Σε 79 χώρες χρησιμοποιείται. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα προβολή της Ένωσης. Πολλές φορές ο ΙΕ ή άλλοι οργανισμοί βάζουν το λογότυπό τους, αλλά όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά και σε ό,τι αφορά την προβολή των αξιών της Ένωσης, όλες τις μορφές αναπτυξιακής βοήθειας. Θα επανέλθω στο πλαίσιο της συζήτησης. Τα λέω γρήγορα τώρα, γιατί μπορείτε να τα διαβάσετε και στην έκθεση, για την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ε, ή αναπτυξιακούς οργανισμούς ε, της Ένωσης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Τι θέλουμε, να υπάρχει έλεγχο των έργων, εσωτερική έλεγχη και να υπάρχει και ρήτρα σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει επίσης ευρωπαϊκή δημοσιονομική στήριξη, κίνδυνοι και προκλήσεις ε, για το ΦΕΔ και να προσέξουμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή έτσι, εκτροπή. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, αλλά βλέπουμε ότι μπαίνει πολύ ε, μεγάλη έμφαση και δίνονται πολλά κονδύλια για κάτι που δεν είναι προτεραιότητα στο ΕΤΑ, δηλαδή την ασφάλεια. Τώρα για το καταπίστευμα για την Αφρική. Υπάρχουν πολλά θέματα ε, σε ό,τι αφορά την προστέμενη αξία αυτού του ταμείου και ζητούμε η Κομισιόν να εγγυηθεί ιδίω πώ δεν θα πρέπει να υπερτερεί η, η παράμετρος της ασφάλειας από τις ανάγκες των δικαιούχων χωρών. Δεν θέλουμε να χρηματοδοτούνται προγράμματα τα οποία εφαρμόζουν τοπικές κρατικές αρχές όπως ε, ξέρετε τι έγινε με τη Λιβύη. Είχαμε πολύ μεγάλες επικρίσεις για το, ε, για το Σουδάν ε, που έχουμε παρεμβάσει των δικαιωμάτων. Και υπάρχει μια παράγραφος για τον Ήγηρα και την Ερυθρέα. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα σταματήσω λίγο για την Ερυθρέα γιατί έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Θα σας τα πω εν συντομία. Τον Απρίλιο του 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του καταπιστεύοντος για την Αφρική άρχισε να υποστηρίζει τον αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο ενός έργου για την αποκατάσταση του βασικού δικού δικτύου στην Ερυθρέα που στόχο επισήμως είχε να υπάρξει σύνδεση με το λιμάνι. 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κονδύλι. Πρώτη, φορά, ε, πρώτη φάση γνώμη, ε, του έργου. Τι λένε οι τεχνικές προδιαγραφές. 20 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ένωση και εκχωρήθηκε ε, στο ΙΝΟΨΑ από τον ΟΗΕ μια οργάνωση που θα αναλάμβανε. Και η αρμόδια εταιρεία από την Ερυθρέα θα έκανε ένα διαγωνισμό, ε, για, μάλλον θα προσέφευγε ε, στο εργατικό δυναμικό, εκεί, που μιλάμε για καταναγκαστική εργασία. Εκεί υπάρχει στατιωτική θητεία, είναι οι έφεδροι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν. Ε, ουσιαστικά πρόκειται για καταναγκαστική εργασία, γιατί έχουμε δικτατορία στην Ερυθρέα. Ε, ήρθαν ε, υπόψη μας αυτά ε, τα θέματα και κατέθεσα δύο προφορικές ερωτήσεις στην Κομισιόν. Η μία αφορούσε στο συγκεκριμένο έργο, η δεύτερη το θέμα της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας από το καθεστώς. Και η πρώτη ερώτηση είναι πως η Κομισιόν υπέγραψε μία σύμβαση που αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει εργατικό δυναμικό από τις εθνικές υπηρεσίες, δηλαδή ε, ουσιαστικά ε, θα αναγκάσει τον κόσμο να εργάζεται αυτούς τους ε, ανθρώπους που κάνουν στρατιωτική θητεία. Δεν έχω ε, καμία απάντηση. Στη δεύτερη περίπτωση, 28 Νοεμβρίου 2018, είχαμε μια ακρόαση και έθεσα στον Επίτροπο Μίμητσα ε, την ερώτηση. Όταν συζητούσαμε την απαλλαγή 18 για τα ταμεία. Διακόπτεται η ομιλήτρια. Ποιος σε προεδρεύει, γιατί δεν υπάρχει κανένας πάνω στο βήμα. Είναι σημαντικό όμως, γιατί σίγουρα θα δεχθώ ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Χολμάγερ, με υποστήριξε, γιατί στο ερώτημα αν η Ένωση είναι κάπως τελικά συνένοχη αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ που δίνει για το δικό δίκτυο αλλά τελικά ε, δείχνει ε, σαν να στηρίζει το καταναγκαστικό, την καταναγκαστική εργασία. Καμία απάντηση από τον κύριο Μίμητσα, γι' αυτό και η κυρία Χολμάιερ το ξαναέθεσε το διόρθωμα. Πάλι δεν πήραμε απάντηση. Τι πήραμε όμως τελικά, πήραμε γραπτή απάντηση από τη γραμματεία της Επιτροπής Κόντ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί η Ένωση, λέει, να είναι υπεύθυνη για την παραβίαση, παραβίαση των δικαιωμάτων. Δεν το διαχειριστάμε σε αυτό το έργο. Έχει εκχωρήσει στο Ίνοψ την, ε, ε, ανά, την παρακολούθηση του έργου αυτού. Ουσιαστικά χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η αρμόδια εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα παρακολουθεί για να γίνονται σεβαστοί κανόνες κτλ. κτλ. Ήδη πρόκειται κάτι απαράδεκτο. Μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια. Χρησιμοποιούμε μία οργάνωση του ΟΗΕ για την εκτέλεση του έργου, αλλά λέμε εμείς πλέον ανήπτουμε τα μας. Δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Απ' την άλλη πλευρά, υπήρξε ένα άρθρο στη New York Times 8 Ιανουαρίου του 2020. Τι μαθαίνουμε, ότι η ΝΟΠΣ αυτό το γραφείο λέει δεν έχουμε ε, γραφεία στην Ερυθρέα και δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Έγιναν δύο-τρεις συναντήσεις επιτόπου, αλλά ουσιαστικά από την αιγίδα της κυβέρνησης Ερυθρέας. Και τι άλλο μαθαίνουμε τελικά, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν εγώ είχα θέσει το ερώτημα και πέρματα την γραπτή απάντηση, η Κομισιόν έδωσε άλλα 60 εκατομμύρια, δεύτερη δόση. 14 Γενάρη, τώρα παίρνω την επίσημη απάντηση στην προφορική μου ερώτηση εκ μέρους της νέας επιτρόπου που μου δίνει ακριβώ την ίδια ε, ψευδή απάντηση, δηλαδή ότι ο οργανισμός του ΟΗΕ είναι αρμόδιος, ενώ ήδη από το ενόψη είχαμε γραπτή διάψευση, γραπτό έγγραφο από το ενόψη που λέει ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Και αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Α, ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Χολμάκη. Η νέα επίτροπος μάλλον δεν παίρνει σωστές συμβουλές, ε, ούτε την ενημερώνει σωστά ή δεν δίνει αυτή όλες τις πληροφορίες. Και πιστεύω ότι έχουμε εδώ ένα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα εμείς οι ευρωβουλευτές. Γιατί σας τα λέω όμως όλα αυτά. Πρώτον, κάνει αυτή την πολύ πλήρη έρευνα η εφημερίδα New York Times. Δεύτερον, η Κομισιόν δίνει χρήματα στην Ερυθρέα χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς κανένα όρο. Τρίτον, η Κομισιόν μας απαντάει η ΝΟΠΣ, ε, αυτό, αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ ελέγχει, όμως σε γραπτή απάντηση η ΝΟΠΣ λέει δεν ελέγχουμε. Άρα, αυτή τη στιγμή η ΜΚΟ επιτίθενται. Ε, θα έχουμε και καταγγελία, προσφυγή στο δικαστήριο που λέει ότι η Κομισιόν κατά κάποιο τρόπο ε, στηρίζει, χρηματοδοτητή την καταναγκαστική εργασία. Και εμείς δεν είχαμε καμία πρόσβαση εκ των προτέρων. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτού του είδους τα έργα, γιατί αποφάσισαν τα κράτη, όχι το κοινοβούλιο. Άρα μας βάζουν και εμά το ίδιο το καζάνι. Και αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί αν δεν κάνουμε τίποτα, όλες οι ΜΚΟ θα μας επιτεθούν λέγοντα: ορίστε να τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτεί μια δικτατορία στο πρόσωπο της Ερυθρέας. Γιατί φτιάχνουμε ένα δρόμο από την Αιθιοπία μέχρι τα λιμάνια της Ερυθρέας. Αλλά αυτό πιο ωφελεί. Άμα το σκαλίσουμε λίγο παραπάνω, θα σας πω, εγώ ας πούμε που είμαι από την Ερυθρέα, βλέπω ότι η κυβέρνησή μου έχει χρήματα για να φτιάχνει δρόμους και λέω τέλεια, καταπληκτικά. Θα τη στηρίξω την κυβέρνηση αυτή, που όμως είναι δικτατορία. Και η Κομισιόν δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, κανένα στάθμισμα. Και δεν ε, φρόντισε ούτε καν να υπάρξει ένας αποτελεσματικός έλεγχος. Εγώ θέλω να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αν συμφωνείτε, θα πρέπει να πούμε στην Κομισιόν ότι περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και γι' αυτό και αναβάλουμε τη χωρίς απαλλαγή για έξι μήνες. Έχετε έξι μήνες δηλαδή Κομισιόν για να μας δώσετε απαντήσεις, ώστε εμείς ως ευρωβουλευτές να μπορέσουμε μετά να δικαιολογηθούμε ε, απέναντι στην κοινή γνώμη. Αλλά εμείς θα είμαστε αντικείμενο επίθεσης. Είναι η πρώτη φορά, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, ε, δεν δίνονται μόνο 20 εκατομμύρια, δόθηκαν και άλλα 60. Και μας κορόιδεψαν. Γιατί κυρία Πρόεδρε, όταν είχαμε την ακρόαση με τον κύριο Μίμητσα, δεν μας το είπε ότι θα ξανά δίνουν λεφτά, θα δίνανε 60 εκατομμύρια επιπλέον. Άρα θέλουμε ε, τις πληροφορίες που δεν μας δώσανε, δεν μας είπαν για την καταναγκαστική εργασία. Μας δίνουν ψευδείς πληροφορίες, μας λένε το ΙΝΟΨ ελέγχει, ενώ το λέει δεν ελέγχει τίποτα και μετά μα λένε αν ναι, είναι σημαντικό γιατί πρέπει να έχουμε πρόσβαση στη χώρα. Ναι, να έχουμε πρόσβαση, αλλά για να βοηθήσουμε στον τομέα τη παιδεία και τη υγεία. Όχι για το δικό δίκτυο. Τι νόημα έχει. Ποιο θα ωφεληθεί, η Αιθιοπία θα ωφεληθεί. Γιατί οι Ερυθρέοι ουσιαστικά ε, το μόνο που κάνουν ότι τελικά ε, ωφελείται η κυβέρνηση γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι κάνει έργο η κυβέρνηση που είναι μια δικτατορία. Προσέξτε πολύ όμως, γιατί θα μας ε, ε, εξαπολύσουν ε, δρυμία επίθεση. Εμείς πρέπει να το πούμε ως Ευρωβουλευτές. Δεν συμφωνούμε. Δεν ξέρω τι πιστεύει και η Πρόεδρος, αλλά μας έχουν βάλει σε πολύ δύσκολη θέση. Πολύ λεπτή θέση. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας επιστήσω την προσοχή ότι, στο ότι στη δική μου έκθεση ασχολήθηκα με αυτό και αναφέρω ότι δεν προβλέπεται κάποια δυνατότητα, οποιαδήποτε περίπτωση καταναγκαστικής εργασίας, δουλείας, οποιαδήποτε μορφή δουλείας να σχετίζεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το αναφέρω αυτό. Η χρηματοδότηση της καταναγκαστικής εργασίας είναι τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό έχω καλέσει και τα, τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να λάβουν θέση Το Διεθνές Δικαστήριο ασχολείται με αυτό εδώ και πάρα πολλά. Το, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ελεκτικό Συνέδριο, με συγχωρείτε, ασχολείται με αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζητά να δοθεί μία λύση και πρέπει να ασκηθούν πιέσεις. Και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω προσθέσει και εγώ κάποια σημεία στην έκθεσή μου, τα οποία συζητήσαμε, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Ντάβιντ Λέγκα, σκιώδη συγητή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την ε, καλογραμμένη έκθεση. Νομίζω πως η δομή της είναι λογικότατη, είναι κατανοητή, περιέχει συγκεκριμένα στα ε, στοιχεία και ασχολείται με τα αυξανόμενα ποσοστά σφάλματος ε, για παράδειγμα την ε, αδυναμία συμμόρφωσης σε ό,τι φορά τις δημόσιες προμήθειες και άλλα. Έχετε τονίσει στην έκθεσή σας τα σημεία που με απασχολούν και εμένα περισσότερο από όλα. η ανεπαρκής έλλειψη μάλλον η αναπαρκής ύπαρξη συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και οι ανησυχίες ε, που προκύπτουν σχετικά με το που πάνε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που συμπεριλάβατε τα στοιχεία αυτά στην έκθεσή σας, καθώς και για το ότι δίνετε έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην έκθεση τονίζεται η ορατότητα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσπιση του κράτους ε, δικαίου. Επίσης, τονίζεται και ε, το κράτος δικαίου ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ε, κάνω και μία πρόταση στην έκθεση να μειωθεί η έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, διότι δεν είναι αυτός ο στόχος ε, της ε, έκθεσης. Ε, στόχος μας θα πρέπει να είναι η διατήρηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και σωστά το είπατε κι εσείς, υπάρχει ο κίνδυνος να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα και να απομακρυνθούμε τον αρχικό μας στόχο που είναι η απαλήφη της φτώχειας. Τώρα σε ό,τι αφορά τα σχόλια για την Ερυθρέα και την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με την ε, χρήση των ε, Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, εγώ να σας πω πως δεν προτίθεμαι να δώσω απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτού μας ξεκαθαρίσει πού χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα και αν όντω υπήρξε καταναγκαστική εργασία χρηματοδοτούμενη με ευρωπαϊκά κονδύλια. Χρειαζόμαστε απαντήσεις λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και τίνω και εγώ προ ε, το να ζητήσω αναβολή πρωτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Αναρωτιέμαι όμω γιατί έχετε προτείνει το Σεπτέμβριο. Εγώ θα ήθελα απαντήσει στο συντομότερο και ο Σεπτέμβριο μου φαίνεται μακριά. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τότε. Και κάτι άλλο. Σε γενικέ γραμμέ νομίζω πω ε, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πιο δυνατή γλώσσα. Δεν μπορούμε να σημειώνουμε απλά ότι ε, αυτή τη στιγμή τρέχουν 19 διαφορετικές έρευνες. Δεν μπορούμε να λέμε σημειώνουμε ότι. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ισχυρότερη γλώσσα, περισσότερη έμφαση, έμφαση στην απαλυφή της ευτόχειας, λιγότερη έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα για τους λόγους που σας ανέφερα και να επαναλάβω στα εισαγωγικά σε ό,τι, ό,τι είπατε και εσείς ε, στην δική σας έκθεση ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για καταναγκαστική εργασία στην Ερυθρέα και να φροντίσουμε να δώσουμε την δέουσα έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πένκοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή που παρουσίασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Στο σχέδιο της έκθεσης καλύπτονται οι σημαντικότερες πτυχές του ζητήματος και χαιρετίζουμε το ότι πολλές από τις δικές μας παρατηρήσεις και ιδέες τις έχετε λάβει υπόψη σας στην έκθεσή σας. Αυτό το εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος. Παράλληλα βέβαια έχουμε την εντύπωση ότι η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτεύγματα και βέβαια χαιρόμαστε για το ότι επικρίνει τους τομείς εκείνους όπου θα πρέπει να έχουμε περισσότερη βελτίωση όπως η βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι στην έκθεσή σας λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να έχει πιο συστηματική στάση απέναντι στη διαφάνεια και τη λογοδοσία για τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και εστιάζεστε βέβαια και εσείς στο βασικό στόχο που είναι η μείωση της φτώχειας. Η έκθεση αναφέρεται επίση στι ανησυχίε που έχουμε όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει την χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη. Καταλήγεται στο συμπέρασμα δεν θα υπάρξει τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα. Και όπω είπε και ο κύριο Λέγκα πριν από λίγο, και εμεί ανησυχούμε για το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματος, το, οποίο αυξάνεται για δεύτερο συνεχές έτος και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να ανατρέψει την τάση αυτή. Όσον αφορά τώρα τις συστάσεις σας, θα πρέπει σε αυτές να συμπεριλάβετε μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία θα πρέπει να λάβει πιο κατάλληλα μέτρα και να χρησιμοποιήσει καλύτερα μέσα τα οποία θα πρέπει να τα εξηγεί καλύτερα και να τα διαθέτει στις τρίτες χώρες. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί κάπου στην έκθεσή σας. Και βέβαια να αναφερθώ και στο ζήτημα αυτό, το οποίο θίξατε και εσείς εκτενέστατα ε, εισηγήτρια. Χρειαζόμαστε σαφώς περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα της Ερυθρέας προκειμένου να καταφέρουμε και εμείς να αποφανθούμε οριστικά. Αυτή τη στιγμή μας δοθούν βέβαια περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολιβιέ Σαστέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με την σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ριβαζή, την εισηγήτριά μας για την εργασία της και να ευχαριστήσω βέβαια και την Επιτροπή μας για την εργασία που έχει επιτελέσει. Εν γέννη συμφωνώ με τους βασικούς προσανατολισμούς του σχεδίου αυτού έκθεσης που με πολύ ωραίο τρόπο παρουσίασε πριν από λίγο η κυρία Ριβαζή. Επιτρέψτε μου να επιμείνω σε τρία σημεία. Δεν θα σας κάνει εντύπωση κυρία Πρόεδρε, διότι τα σημεία αυτά τα ανέφερα και στην συζήτηση απαλλαγής που κάναμε για την Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ψηφιοποίηση, στην, στα δύο φύλλα και στην αποτελεσματικότητα στις επιδόσεις καταρχάς. Περισσότερους δείκτες επιδόσεων νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δαπανούμε κάθε χρόνο στα πλαίσια των Ταμείων Ανάπτυξης και δεν καταφέρνουμε κάθε φορά να έχουμε τους απαραίτητους δείκτες για να δούμε τελικά αν όντω η δική μας η επέμβαση, η δράση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να χαρτογραφήσουμε περισσότερο τη δραστηριότητά μας και τα προγράμματά μας σε σχέση με τα δύο φύλλα. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μέσω των προγραμμάτων μας μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τις γυναίκες, τα κορίτσια, αν δίνουμε την απαραίτητη έμφαση στα σεξουαλικά ή αναπαραγωγικά δικαιώματα, καταλαβαίνετε ότι κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό να αγνοεί το 50% του πληθυσμού στις χώρες όπου αποτείνεται το πρόγραμμα αυτό. Τρίτον, όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τα μεμονωμένα άτομα, καθώς επίσης και με τους θεσμούς δημοσιού και ιδιωτικούς, στους οποίους απευθυνόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτό το οποίο έχουμε προωθήσει πάρα πολύ τελευταία χρόνια, το more is more ανταυτού νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να αφουγκραστούμε τις πραγματικές ανάγκες των κρατών δικαιούχων και να καταφέρουμε τελικά να προσαρμόσουμε την ενίσχυσή μας στις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται προκειμένου να καταρτιστούν δημοκρατικοί θεσμοί στις χώρες δικαιούχους. Όσον αφορά τώρα την Ερυθρέα, αυτό το οποίο μάθαμε πρόσφατα για τη χώρα αυτή βέβαια μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και απογοήτευση. Νομίζω ότι ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τα σχετικά κονδύλια θα πρέπει να συμβάλλουν στην πρόθεση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και στη θέσπιση ενός πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε ακόμα όμως τι γίνεται σε σχέση με αυτό. Και αυτό το οποίο βλέπουμε επί του παρόντος είναι ότι ε, δεν θα πρέπει εμεί να αποφασίσουμε ευθύ αμέσω για το αν θα πρέπει να χορηγηθεί ή όχι μια απαλλαγή. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε άμεσα είναι μια έκθεση εμπεριστατωμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποία να έρθει να συμπληρώσει τα στοιχεία τα οποία μα έχει δώσει μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφασίσουμε εμεί εκ των υστέρων αν θα χορηγήσουμε ή όχι απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ, Ολιβιέ. Θα ήθελε κάποιο άλλο το λόγο. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ναι, πρώτα θα λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς στη συνέχεια. Πώς θέλετε, θέλετε τώρα, όπως θέλετε. κύριε Ζητόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα τα πω λοιπόν στα αγγλικά. Θα ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση σε κάποια άλλα project των Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπατε και εσείς, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε σωστές πληροφορίες τώρα και όχι σε 6 μήνες. Με σόκαρε το άρθρο του New York Times. Και μετά ακούω ότι εσείς ζητάτε να μας δώσουν πληροφορίες έξι μήνες αργότερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε την εξήγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πρόκειται για τα δικά μα χρήματα και θέλουμε να ξέρουμε πού πηγαίνουν. Και εγώ δεν θέλω να δίνω χρήματα σε καταναγκαστική εργασία, σε δουλεία. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, πως στην Ερυθρέα υπάρχει δικτατορία, γι' αυτό και είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες. και συμφωνώ απόλυτα με τον σκιοδησηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Λέγκα, ο οποίος είπε πράγματα με τα οποία είμαι απόλυτα σύμφωνος. Η έκθεση θα πρέπει να εστιάσει σε θέματα ανάπτυξης. αλλά και στα σχετικά με αυτή. η κυρία Χολμάιερ επίσης ήταν σε μία αποστολή το 2015 ή 2016, αν δεν κάνω λάθος, στο Λίβανο. σε συνεργασία με ένα project από την UNRVA. Είναι μια οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες ε, στην Παλαιστίνη. Και πραγματικά ήταν απίστευτο αυτό που ακούσαμε, ότι δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο, δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τα πάντα, πού πάνε τα χρήματα. Εμείς τους, ζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε δράσεις ριζοσπαστικοποίησης και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και μετά μας είπαν ότι όχι, ναι, ξέρετε, πάνε σε, σε μια άλλη παλαιστινιακή οργάνωση, και μετά χάνουμε λίγο την επισκόπηση. Και υπήρχαν προβλήματα και με το γραφείο διασύνδεσης ε, στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Ήταν λοιπόν επονίδιστο αυτό. Δηλαδή, να πείστε αυτό πώς μας εξήγησαν τι συμβαίνει και τι απάντησαν στις κατηγορίες μας. Ε, μας είπαν χρειάζεται να μας εμπιστευτείτε. Είμαστε Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και Εξορισμού δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Και αυτή είναι η θέση μας. Και εγώ ονομάζομαι Θωμάς, είμαι άπιστος, εκγενετής. Χρειάζεται πρώτα λοιπόν να ζητήσουμε μια επίσημη απάντηση από τα Ηνωμένα Έθνη, μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έπειτα θα δώσουμε ή όχι την απαλλαγή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πέξα, έπειτα και Πινιαντόλη και είστε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, σύντομα. Μια παρατήρηση για τη διαδικασία. Άνθρωποι είμαστε και δεν πρέπει να φύγω εγώ, αλλά όταν έχουμε επίσημη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής, ε, θέλω να σας παρακαλέσω αν ε, φεύγετε είτε να διακόπτετε τη συνεδρίαση είτε να επιφορτίσετε κάποιον άλλο ε, να προεδρεύσει απουσία σας. Να μην συμβεί αυτό όταν έχουμε μια επίσημη συνεδρίαση. Αλλά αν δεν είναι κανείς εδώ αντιπρόεδρος και πρέπει να πάω για πέντε λεπτά στην τουαλέτα, κύριε Πέξα, τι να κάνω. Να σας κάνω να περιμένετε όλοι γιατί πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Δεν θεωρώ πια ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει αν δεν είμαι εγώ παρούσα. Ε, δεν είμαι πια και τόσο σημαντική και αναντικατάστατη και νομίζω ότι η ε, κυρία Ριβαζή που ξέρω και την άποψή της και το περιεχόμενο της έκθεσης ε, και την στηρίζω νομίζω ότι το άντεξε τέλος πάντων ε, αφού δυστυχώς δεν είναι κανένας αντιπρόεδρος εδώ σήμερα να μην το παίρνουμε και τόσο σοβαρά η συνάδελφος πίνει αντόλη θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Συγήτρια, για την έκθεσή σας αυτή και κυρίως διότι αποφασίστατε να εστιαστείτε σε αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ερυθρέα για την δημιουργία του δρόμου αυτού. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ σημαντική, καταρχάς όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έλεγχη όμω είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε πώ κατασκευάζεται αυτό ο δρόμο να σας πω ποια είναι η Ιταλική εμπειρία. Στην Σομαλία κατασκευάστηκε ένας δρόμος και ο δρόμος αυτό κατασκευάστηκε κυρίως ε, για να αποθηκευτούν τελικά κάποια απορρίμματα στο υπέδαφος τελικά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε από τεχνικής πλευράς πώς κατασκευάζεται ο δρόμος. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει το πολύ ευχάριστο έργο να απαντήσει η Κομισιόν στις δύσκολες ερωτήσεις. Λίκ Πάγιο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω στο σύνολο των σχολείων και των ερωτήσεων δεδομένου του περιορισμένου χρόνου. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ριβαζή, για την έκθεσή της και την επικοδομητική της προσέγγιση. Να ευχαριστήσω και το Ελληνικτικό Συνέδριο για την έκθεσή του για το 2018. Όπως ε, κάθε χρονιά, έτσι και φέτος λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελληνικτικού Συνεδρίου για την ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όπως ε, κάνουμε κάθε χρόνο μέσω των ε, σχεδίων δράσης μας. Στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σημειώνεται ότι υπάρχει αύξηση των ποσοστών ασφάλματος, κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μεταξύ του 2, μάλλον είναι μεταξύ του 1,2 και το 9,1. 1,2 είναι η βάση και 9,1 είναι το η ανώτατη τιμή και μέσα σε, αυτές τη, σε αυτή την περιοχή τιμών κυμαίνονται τα σφάλματα που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μεταξύ του 2017 και του 2018 είχαμε επιδείνωση ό,τι αφορά τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Πόσο μάλλον που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εξολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και ξέρετε ότι έχουμε ένα σύστημα υπολογισμού των ποσοστών σφάλματο, που δεν είναι το ίδιο με αυτό το ελεγκτικό συνεδρίο γιατί ο στόχος μας είναι διαφορετικός σε σχέση με το ελεγκτικό συνεδρίο. Εμεί θέλουμε συμπληρωματικέ πληροφορίες να δώσουμε. Το ελεγκτικό συνεδρίο μετράει τις δραστηριότητες του έτους ε, και εμείς το σύνολο των συμβάσεων που ολοκληρώθηκαν στη δέκα τη χρονιά. ανεξαρτήτως έτου και έτσι μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου άπαξ και εκτελέστηκαν όλοι οι εσωτερικοί έλεγχοι και εκεί βασίζουμε το ποσοστό σφάλματος. Στη δική μας περίπτωση βλέπουμε συνεχή μείωση του ποσοστού σφάλματος ε, λόγω και των διαφόρων σχεδίων δράση μα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ε, να διορθώνει τα πράγματα από τη στιγμή που έχει γίνει η πληρωμή και μέχρι τη στιγμή που κλείνει, ολοκληρώνεται ένα έργο. Βλέπουμε ακόμη και σημειώνουμε τις ανησυχίες σας ό,τι αφορά τους διεθνείς οργανισμούς, είτε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα, την ε, διαφάνεια, τον έλεγχο, των δραστηριοτήτων, τον λογιστικό έλεγχο κτλ. Ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας. Επίσης, ε, στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου δίνεται έμφαση στην πρόσβαση στα έγγραφα, κάτι που υπονοεί ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει, πρόβλημα υπάρχει, αλλά οι διεθνείς οργανισμοί στο ποσοστό σφάλματος ε, αντιπροσωπεύονται στο ε, πεδίο που τους αναλογεί. Δεν υπάρχει υπερεκπροσώπησή τους, δηλαδή στο ποσοστό σφάλματος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυξάνουμε και τις πιέσεις μας, ώστε να παρέχεται στις ελεγκτικές αρχές έγκαιρα ε, το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων. Αν είχε δοθεί εγκαίρως ε, η τεκμηρίωση, ε, δεν θα είχε γίνει μηδενικό το σφάλμα, αλλά σίγουρα βοηθάει. Το λέει και το Ελληνικό Συνέδριο. Αυτό ό,τι αφορά τι ε, παρατηρήσει τώρα. Για τι μεσονομικέ παρατηρήσει, τη μεσονομική στήριξη. Εδώ και 25 χρόνια παρέχουμε αυτή την υποστήριξη. Ε, θέλουμε να σέβεται την αρχή της ευθυγράμμισης με τις ε, αναπτυξιακές πολιτικές ε, για να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες εταίρους να εφαρμόσουν πολιτικές υπέρ της εκρίζωσης της στόχιας και όχι να παρακάπτουν το σύστημα. Θέλουμε επίσης μεγαλύτερη επιτήρηση από τις ελληνικές αρχές των κρατών εταίρων είτε είναι το οικονομικό, είτε είναι το ελληνικό συνέδριο, είτε είναι εσωτερικό ελεγκτής. Έχουμε βελτιωθεί όλα αυτά τα 25 χρόνια. Σίγουρα πρέπει βέβαια να υπάρχει συγκεκριμένα παρακολούθηση της μεσονομικής στήριξης. Ε, υπάρχουν εκθέσεις και εκτιμήσεις που δείχνουν συσχέτιση και αντιστοιχεία μεταξύ των προγραμμάτων διασυνομικής στήριξης και της αποτρεσματικότητας των δράσεών μας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Και φτάνω τώρα στο θέμα της ημέρας, την Ερυθρέα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο χρόνο για να σας εξηγήσω το υπόβαθρο. Το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα της Ερυθρέας εγκρίθηκε νομίζω το 2015, δηλαδή ε, στην αρχή του χρηματοοικονομικού αυτού κύκλου. Εγκρίθηκε μετά τη γνωμοδότηση των κρατών μελών και μετά και ε, το στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη από την αρχή Επομένως υπήρχε ένα έγγραφο που ήταν αντικείμενο συνένεσης. Όταν τώρα ε, ξεκίνησε εκ νέου η συνεργασία μας με την Ερυθρέα το 2019, λάβαμε την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη από την Διαχειριστική Επιτροπή, όπου προσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη, ξεκίνησε διάλογος με την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε έγκριση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου, αλλά υπήρξε διάλογος, υπήρξε μια συνεννόηση. Ποιο είναι το πλαίσιο τώρα. Έχουμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ερυθρέας και Αιθιοπίας, μια συμφωνία ειρηνευτική. Ο Αμπί Χαμέντο, ο και βραβευμένος με Νόμπελ, ξανά ε, ζητά ε, να υπάρξει επαφή και ειρήνευση με την Ερυθρέα. Απ' την άλλη έχουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που αναστέλει τις κυρώσεις και το εμπάργκο όπλων και όλοι οι φορείς δραστηριοποιούνται για να εργαστούν στην Ερυθρέα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν φυσικά και καταδικάζει κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα Λυπούμαστε που υπάρχει αυτή η στρατιωτική θητεία μέχρι και τα 40 χρόνια, ε, δηλαδή δεν είναι πια νέοι, αλλά εξακολουθούν να υπηρετούν ε, οι ε, άντρες εκεί. Σίγουρα χρειάζονται ρυθμίσει. Δεύτερον, μάλλον τρίτον, σε καμιά περίπτωση τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν στηρίζουν το σύστημα της καταναγκαστικής εργασίας. Ούτε ένα ευρώ δεν πηγαίνει για αυτή τη δουλειά. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό το έργο, δεν είναι ανέγερση ε, οδικού, μάλλον αυτοκινητόδρομου αλλά αποκατάσταση, αποκατάσταση του οδικού δικτύου, του συγκεκριμένου αυτοκινητοδρόμου. Και παρέχουμε εξοπλισμό. Δεν χρηματοδοτούμε το σύστημα. Τούτου λεχθέντος αυτό το σύστημα με τη θητεία ε, είναι ένα γενικευμένο σύστημα στην ΕΦΤΑ, δηλαδή ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο παρεμβαίνουμε, είτε είναι ο τομέα της υγεία, είναι ο τομέα ή τη αποκατάσταση του οδικού δικτύου, έχουμε να κάνουμε ακριβώ με αυτό το σύστημα που χρησιμοποιεί ε, τους ε, εφέδρους, τους στρατιώτες για να εκτελούν τι εργασίε αυτές εκ μέρου της κυβέρνηση. Άρα τελικά ποιο είναι το θέμα που τίθεται. Θέλουμε να είμαστε παρόντες σε αυτή τη χώρα και υπό ποιους όρους ή όχι. Ο πολιτικός προσανατολισμός του 2019 σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη είναι να είμαστε παρόντες στη χώρα. Βεβαίως πάντοτε όντας ιδιαίτερα επικριτική απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην Ερυθρέα. Δεν υπάρχει υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κομισιόν σε καμία περίπτωση σε ένα σύστημα δουλείας ε, ή καταναγκαστικής εργασίας. Ακόμη και αν αναγνωρίζουμε ότι το σύστημα καταναγκαστικής εργασίας υπάρχει και υπάρχει σε όλους τους τομείς δραστηριότητας στη χώρα αυτή. Τώρα, για την ΕΝΟΠΣ, αυτή την υπηρεσία του ΟΗΕ. Το άρθρο του New York Times ε, τέλος πάντων ε, οι δηλώσεις που γίνονται από αυτή την, από αυτή την υπηρεσία είναι πάρα πολύ αδέξιες και λυπούμαστε γι' αυτό. Δεν δεσμευόμαστε, μας δεσμεύουν αυτά που λέει η ΝΟΠΣ ως Κομισιόν. Εμείς αμέσως ξεκινήσαμε με διάλογο με την ΝΟΠΣ και πήραμε πληροφορίες οι οποίες μας επιτρέπουν να πούμε πως η ΝΟΠΣ στους New York Times λέει ότι δεν παρακολουθεί το σύνολο του προγράμματος υποκατάσταση στο δικό αλλά παρακολούθηση συγκεκριμένη υπάρχει για το δικό μας το πρόγραμμα. Είναι κύριος του έργου ο και εμείς παρακολουθούμε τις εργασίες. Επίσης έχουμε ε, στην Ασμάρα αντιπροσωπεία, άρα είμαστε επιτόπου εκεί ή έχουμε παρουσία. Η απαντήση Κομισιόν κομισιων θεωρειται ότι δεν είναι επαρκής. Το σημειώνω. Οι απαντήσεις μας δεν σας ικανοποιούν. Το σημειώνω. Και φυσικά και δεσμεύομαι ότι θα σας δώσουμε το συντομότερο δυνατό απαντήσεις. Δεν μπορώ βέβαια εγώ να ε, μιλήσω για την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής. Είναι δική σας η απόφαση. Αλλά πριν τις 29 Γενάρη, δηλαδή πριν τη στιγμή που θα συζητήσετε τις τροπολογίες, νομίζω τουλάχιστον, θα μπορούμε να σας έχουμε στείλει ε, τις πληροφορίες ε, και ένα έγγραφο που θα περιλαμβάνει τις συμπροματικές αυτές πληροφορίες που σας είπα, που μου ζητήσατε. Δεσμεύουμε επίσης, γιατί όχι, να οργανώσουμε και μια επιτόπια επίσκεψη κοινή Επιτροπών Κοντ και Ντέβε στην Ασμάρα για να δούμε το έργο αυτό. Με τα χαρά σε την προσωπία μας θα το οργανώσει αυτό το ταξίδι, ώστε να δει τη διεισόμαση την κατάσταση εκεί, πώς εκτελείστε το έργο, να έχετε και διάλογο με τις αρχές της χώρας. Άρα, Έχετε εδώ αυτά που σας είπα, είναι εδώ και ο αρμόδιος ε, συνάδελφος για το κέρας της Αφρικής. Έχετε τη δέσμευσή μας, θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν ως βουλευτές να μπορέσετε να διενεργήσετε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και δράσεων της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ωραία, θα ήθελα να τοποθετηθώ και εγώ για αυτό που ακούστηκε, τους έξι μήνες. Οι έξι μήνες είναι η μέγιστη προθεσμία, είναι το ανώτατο που μπορούμε να δώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, ελπίζω να κατανοείτε τι σημαίνει αυτό και θα ήμουν ευγνώμων αν πρώτα το σκεφτόμασταν και γνωρίζαμε όλες τις πτυχές πριν τοποθετηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη εδώ. Και αυτά έχουν ήδη συζητηθεί στο Στρασβούργο, οπότε να σας το υπενθυμίσω και αυτό. Ε, κυρία Ριβαζή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να απαντήσω καταρχάς στους συναδέλφους. Άκουσα προσεκτικά τα όσα είπατε και όντως θα πρέπει να γίνει η διατύπωση λίγο πιο αυστηρή σε κάποια σημεία της έκθεσης. Και σίγουρα θίγονται και αρκετά περιβαλλοντικά ζητήματα όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ξέρετε ότι θέλουμε να καταφέρουμε να περάσουμε τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη στον κοινοτικό προπολογισμό. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι εκ των υστέρων μόνο λαμβάνουμε τι απαραίτητε πληροφορίε. Και αυτό είναι πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Θα έπρεπε εκ των προτέρων να μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες προτού ξεκινήσουν τα συγκεκριμένα έργα για να μπορούμε και εμείς να τοποθετούμαστε κάθε φορά, την ίδια στιγμή δηλαδή που έχουν τις πληροφορίες αυτές και τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που μας δώσατε, θα σας δώσω και εγώ με τη σειρά μου κάποιες πληροφορίες, γιατί α, μας λένε ότι όλα γίνανε μέσω διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε μπλακεί και εμεί ω ευρωβουλευτέ. Η Επιτροπή Κοντ πάντω έχει μια έκθεση για την απαλλαγή 2017 και λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εκφράζει εκ νέου τους επιφυλάξεις του σε σχέση με την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της έγκρισης του ΦΕΔ για ένα δεικτικό εθνικό πρόγραμμα για την Ερυθρέα. Ήδη λοιπόν από το 2017 σας είχαμε προδοποιήσει για το ζήτημα αυτό. Ήδη από τότε γνωρίζαμε ότι αν επενδύαμε στην Ερυθρέα τρόπον την άθε υποστηρίζαμε στο και έμεσα την καταναστική εργασία. Μην λέτε λοιπόν ότι δεν το είχαμε θίξει παλιότερα το ζήτημα αυτό. Και επικρίνατε το Νόψα το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών. Μα έχουμε μία γραπτή δήλωση του UNOPSA στους New York Times, όπου εξηγούν ότι δεν είχαν την αρμοδιότητα να επιτελέσουν ελέγχους όσον αφορά την επιτέλεση του έργου αυτού στην Ερυθρέα και πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια. Αν πραγματικά συνολικά δίνουμε από ό,τι φαίνεται 80 εκατομμύρια ευρώ, ε, μάλλον θα πρέπει να έχουμε και κάποιε απαιτήσει, έτσι δεν είναι, όσον αφορά του όρου, τι προποθέσει και τον έλεγχο. Ενδεχομένω να μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει επιχειρήσει από την Αιθιοπία και την Ερυθρέα. Αυτή τη στιγμή, μετά όσα μα λέτε, από πολιτική πλευρά τουλάχιστον, μα φέρνετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μου επιτεθούν μη κυβερνητικέ οργανώσει, τι θα του απαντήσω θα μου πούνε ότι δώσατε ως Ευρωπαϊκή Ένωση 80 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσετε τελικά τη στάση που διατηρεί η κυβέρνηση Ερυθρέας απέναντι στην καταναγκαστική εργασία. Πάντως, ε, θα θέλαμε πριν από τις 29 Ιανουαρίου να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνω στους σκιώδεις εισηγητές αυτή τη στιγμή λάβουμε τις απαντήσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεδράσουμε εκ νέου και να δούμε τελικά τι στάση διατηρήσουμε και πώς θα ανταποκριθούμε. Θέλω να διατηρήσω μια στάση εντελώ διαφανή σε σχέση με την πρόταση που έκανε πριν από λίγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, το λέω και σε εσά και στου συναδέλφου θα πρέπει να ζητήσουμε να γίνει μια αποστολή δική μας στην Ερυθρέα. Αυτό θα πρέπει να είναι η πρώτη απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επενδύσαμε χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αποστολή από την Επιτροπή μας στην ΚΟΝΤ και από την ΤΕΒΕ, από κοινού. Ξέρετε ότι και η ΤΕΒΕ έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Από κοινού λοιπόν θα πρέπει δύο επιτροπές να πάνε επί τόπου και να έχουμε απόλυτη ελευθερία. Και σας ζητώ συγγνώμη, δεν εμπιστεύομαι καθόλου τους πρέσβεις μας εκεί δεν τους επιτρέπουμε καν να βγουν από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν στη θάλασσα να πάνε οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν ένα μπάνιο αν θέλουν πολύ ο λόγος. Πρόκειται για μια πραγματική δικτατορία. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε εμείς να πάμε επί τόπου, να έχουμε απόλυτη ελευθερία κινήσεων και να συζητήσουμε πραγματικά με του εργαζομένου. Όταν ζητήσαμε από την UNOPS να μας πει πόσοι εργάζονται, πόσε ώρε την εβδομάδα, πόσο πληρώνονται, δεν μα δόθηκε καμία απάντηση. Περιμένετε από εμά να εγκρίνουμε τη χορήγηση 80 εκατομμυρίων ευρώ χωρί να έχουμε καμία πληροφορία για τι συνθήκε εργασία. Πρέπει να πετήσουμε λοιπόν να διοργανωθεί μια αποστολή δική μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ερυθρέα Κατά αυτόν τον τρόπο θα εμπλουτιστεί περισσότερο και συζήτηση. Λοιπόν, έχω κάνει δύο συγκεκριμένε προτάσει. Περιμένω γρήγορα τη δική σα απάντηση. Απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώ και λέω και στου οικοδησηγητέ ότι αυτή τη στιγμή λάβουμε απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να συνεδράσουμε εκ νέου και να δούμε πώ θα καταφέρουμε να εντρογανώσουμε μία αποστολή στην Ερυθρέα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε και κάποιε συγκεκριμένε απαντήσει από του εκεί εργαζομένου. Θα μιλήσουμε και σήμερα το απόγευμα για τις αποστολές Το δεύτερο μισό του έτους. Έχει ήδη αποφασιστεί να πάμε στην Τινησία. Θα μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε και για δεύτερη αποστολή τότε. Αυτό που είναι δύσκολο να κάνουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν τι θα γίνει με την Ερυθρέα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και δεδομένου του καθεστώτος της Ερυθρέας θα είναι δύσκολη απόφαση. Αυτή η απόφαση λοιπόν είναι στο χέρι των κρατών μελών. Βέβαια, αν δεν τοποθετηθούμε κι εμείς και αν δεν λάβουμε θέση, δεν πρόκειται να βελτιωθεί και τίποτα. Είναι λίγο αδιέξοδο αυτή η κατάσταση. Τι κάνουμε με ένα διεφθαρμένο κράτος. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει το ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα υποστηρίξουμε καταναγκαστική εργασία. αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τα θετικά στοιχεία, τις ε, θετικές ε, δομές στη χώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι εμπόριο, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να τονίσουμε τα θετικά και σε καμία περίπτωση δεν στηρίζουμε λοιπόν την δουλεία. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη φήμη μας. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστούμε πολύ και την Μισελ Ριβαζή για την εξαιρετική δουλειά και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Σας ευχαριστώ όλους και θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το πρωί. Καλά πάμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την απαλλαγή στους οργανισμούς. Ο κύριος Δατσίνσκι θα απαλλαγεί αυτό λίγο πρώτος και στη συνέχεια ο κύριος Λιγκούτκο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε στο, στην απαλλαγή για τους οργανισμούς το 2018. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία όσους συμμετείχατε στην ε, κατάρτιση της έκθεσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Καμίλα Βλουτσίνσκα που κάθεται στα αριστερά μου αλλά και όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ζητήσω από τη στιγμή που ο κύριος Τσαρνέτσκι δυστυχώς ε, λείπει λόγω ασθένειας και δεν είναι εδώ, να χωρίσουμε εγώ και ο κύριος Λεγκούτκο την παρουσίαση στα δύο. Θα παρουσιάσουμε βέβαια και τη δουλειά του συναδέλφου που απουσιάζει. Έχουμε λοιπόν 32 αποκεντρωμένες υπηρεσίες που ε, βρίσκονται στη διαδικασία απαλληγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξετάζουμε λοιπόν την αξιοπιστία των λογαριασμών και των 32 αποκεντρωμένων υπηρεσιών για το 2018. Η... Εκδόθηκε το από Συνέδριο γνώμη με επιφύλαξη τόσο για την νομιμότητα και την κανονικότητα των ε, εσόδων, όσο και για τους ε, λογαριασμούς γενικότερα, εκτός από την ΕΑΣΟ, σε όλους εκτός από την ΕΑΣΟ για θέματα πληρωμών. Όμως ε, στην περίπτωση της ΕΑΣΟ πάντα υπήρχαν αρνητικές, μη θετικές γνώμες. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα, για παράδειγμα ζητείται περισσότερη εναρμόνιση στα θέματα πληροφορικής, ανεξάρτητοι ελεκτές σε ορισμένες υπηρεσίες, θέματα με τις δημόσιες προμήθειες. Έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος ό,τι αφορά το ΣΥΣΠΕΡ 2, το εργαλείο δηλαδή διαχείρισης ε, ε, ανθρώπινου δυναμικού το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς μέχρι τώρα. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με τις δημόσιες ε, προμήθειες, για παράδειγμα ανεπαρκή κριτήρια σε ό,τι αφορά την ε, χορήγηση ενός, ε, μιας σύμβασης. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο ανταγωνιστικές διαδικασίες Χρειάζεται περισσότερες αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Τώρα, οι οικονομίες κλίμακας και οι διοικητικές ε, αρμοδιότητες είναι θέμα που αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης ιδιαίτερα σε υπηρεσίες οι οποίες ασκούν ε, παρόμοια δράση. Όμως ε, δεν έχουμε καταφέρει να αναρμονίσουμε τα ε, κριτήρια. Υπάρχουν λήψεις σε ανάλυση, για παράδειγμα, των δεδομένων της αγοράς. Η ΕΣΜΑ, ας πούμε. Το 2018 έγινε μια δημόσια προκήρυξη για νέα γραφεία. Αυτός ο διαγωνισμός ε, θα γινόταν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία τελικά πήγε στο Παρίσι και δεν ε, υπογράφηκε κοινή σύμβαση. Σε ό,τι αφορά τα γραφεία, ορισμένες φορές ε, δεν μπορούμε να έχουμε οικονομίες κλίμακας γιατί μας ε, λείπουν βασικά στοιχεία. Πολλές φορές επίσης οι υπάλληλοι δεν απασχολούνται με, τις, ε, με κανονικού τύπου συμβάσεις. Αυτό έχουν διαπιστώσει οι λεκτές. και είναι μια περίπτωση την οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, από το 2014 έως 2018 επρόκειτο να γίνουν περικοπές στις τάξης του 5%. Σε πολλές περιπτώσεις οι περικοπές αυτές έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, πολλοί μόνιμοι υπάλληλοι έχουν αντικατασταθεί με συμβασιούχους και υπάρχουν αρκετοί από αυτούς τους έκτακτους ή συμβασιούχους υπαλλήλους. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα χρησιμοποιήθηκε μεσάζοντα εταιρείε ε, έβρεσης ε, ανθρώπινου δυναμικού και εδώ έχουν διαπιστωθεί κάποια θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εξωτερικό προσωπικό θα πρέπει να τηρούμε τις ε, διατάξεις, ε, τις ευρωπαϊκές διατάξεις, αλλά έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στην Πολωνία, όπου δεν εφαρμόζονται τέτοιες, ε, αυτές οι νομικές διατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε εάν έχει νόημα να προσλαμβάνεται εξωτερικό προσωπικό, ενώ ε, μπορούμε να προσλαμβάνουμε επιτόπιο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγονται έλεγχοι και βάσει των ελέγχων αυτών, τον περασμένο Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε ε, κάποιες νέες προτάσεις. Διακόπτη κυρία Χολμάρη. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, διότι δυσκολεύονται πολύ να σας ακολουθήσουν οι δερμηνείς. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν τελείωσα. Συγγνώμη. Οι εσωτερικοί έλεγχοι λοιπόν θα πρέπει να θεσμευτούν από τις ε, αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεγκούτκο για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ήσασταν σύντομο όπω το είπατε. Κύριε Λεγκούτκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς δεν έχουμε σε όλους τους οργανισμούς θέσει οι οποίε να θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητε, που θα πρέπει να διαχειριστούν ιδιαίτερα εμπιστευτικά ζητήματα. Βέβαια, στου οργανισμού που έχουμε τέτοιε θέσει, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που μπορούν να έχουν να κάνουν με κατάχρηση εξουσία. Και δύο οργανισμοί, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων δεν έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένη στρατηγική για να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα που προκύπτουν. Και επίσης υπάρχει και ένας συγκεκριμένος κίνδυνος που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται ε, η κοστολόγηση διαφόρων υπηρεσιών. Και έχουμε εδώ την ΕΣΜΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, το Κέντρο Μετάφρασης, καθώς επίσης και την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Εφτά λοιπόν οργανισμοί, οι οποίοι έχουν ε, έσοδα τα οποία προέρχονται από συγκεκριμένες υπηρεσίες, από κοστολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και πολλές φορές η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την κοστολόγηση μπορεί να είναι παράτυπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι συγκεκριμένοι αυτοί οι οργανισμοί να προσαρμόσουν έτσι τους κανονισμούς τους έτσι ώστε τα τέλη τα οποία χρεώνουν, οι υπηρεσίες οι οποίες κοστολογούν να υπολογίζονται με συγκεκριμένο τρόπο, με τον σωστό τρόπο και όχι με παράτυπο τρόπο. Όσον αφορά τώρα την ΕΑΖΟ, το 2018 το ελεκτικό συνέδριο κατέληξε σε γνώμη με επιφύλαξη όσον αφορά την νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών. Τα αποτελέσματα για τα έτη 2016 και 2017 όμως δεν ήταν θετικά και είχαμε αρνητική γνωμοδότηση από το λεκτικό συνέδριο. Ο λόγος για τον οποίο εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση το λεκτικό συνέδριο έχει να κάνει με σημαντικά σφάλματα που γίνανε σε σχέση με ε, συμβάσεις για την πρόσληψη προσωρινού ε, προσωπικού στην Ελλάδα. Είχαν να κάνουν επίσης με κάποιες παράτυπες συμβάσεις όσον αφορά ε, την ε, οργάνωση ταξιδίων, υπηρεσίες οι οποίες δόθηκαν από το κέντρο, το hotspot στη Λέσβο. Επίσης, στην έκθεση του 2017, του Ελεκτικού Συνεδρίου πάντα για την ΕΑΖΟ, λέγεται ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα όσον αφορά με την νομιμότητα και την κανονικότητα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και ότι υπήρχαν επίσης και πολλές διοικητικές αδυναμίες. Έκτοτε η κατάσταση έχει βελτιωθεί, ορισμένα διορθωτικά μέτρα ελήφθησαν από τα διευθυντικά στελέχη της ΕΑΖΟ και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται τώρα. Η διαδικασία χορήγησης συμβάσεων που χρησιμοποίησε το 2018 η ΑΖΟ και αυτή η διαδικασία πάλι δεν ήταν η πλέον κατάλληλη όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία. Το ελεκτικό συνέδριο τόνισε ότι ε, η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της ΕΑΖΟ επιδεινώθηκε ιδίω κατά την εξέταση της κατάστασης που έγινε το 2017. Τώρα, όσον αφορά το επόμενο έτος, το 2018, είχαμε 278 άτομα προσωπικό και η αύξηση στο προσωπικό πάλι ήταν πολύ χαμηλή το 2018, μολονότι είχαν εντοπιστεί πολλά κενά και 70 θέσεις θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί, οι οποίες όμως παραμείνανε κενές. Και μέχρι τα τέλη του 2018, 4 στις 5 διευθυντικές θέσεις είτε είχαν ανασταλεί είτε ήταν κενές. Ο οργανισμός λοιπόν αυτός βασίζεται πάρα πολύ ακόμα στους πόρους που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, ιδίως όσον αφορά τους αποσπασμένους εμπειρογνώμονες. Και δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων και αυτό το έχουν θίξει πολλές φορές και τα κράτη-μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως τώρα διορθωτικό μέτρο αποφασίστηκε να γίνει μια πρόσληψη τοπικού προσωπικού. Εν γέννη πάντως ε, η πολιτική ανθρωπίνων πόρων που ακολουθείται από την ΕΑΖΟ δεν είναι βέλτιστη και αυτό βέβαια ζημιώνει και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού αυτού. Οι εισηγητέ λοιπόν λένε ότι θα πρέπει να δοθεί απαλλογή σε όλου του οργανισμού με εξαίρεση την ΕΑΖΟ, μολονότι γνωρίζουμε ότι έχει ε, σημειωθεί μια κάποια πρόοδο. Θα θέλαμε την περίπτωση τη ΕΑΖΟ να τη συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα μαζί σα, πρωτοχωρηγήσουμε απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ο σκιώτης συγκεκριτής από το ΕΛΚ παρακαλώ, κύριος Νόβακοφ, Αντρέη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, τον τους και όσους και τους ε, συμβούλους και συνεργάτες μας φυσικά και να ξεκινήσω με μια ιστορία το σχολείο με την απαλλαγή. Δεν συνηθίζεται στην κόντα, αλλά είναι έτσι μια ιστορία που μου αρέσει πολύ και νομίζω ότι έχει και κάποια σχέση με τη σημερινή συνάντηση. Ένας βασιλιάς λοιπόν έχει τρεις ε, γιους και θέλει να κάνει το σοφότερο βασιλιά. Ο πρώτος ε, παίρνει όλα τα όπλα, ο δεύτερος όλο το χρυσό του βασιλείου και ο τρίτος μόνο ζάχαρη και αλάτι. Οι πρώτοι δύο λένε αφού έχουμε όλα τα όπλα και το χρυσό μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε απέναντι στους γείτονες, στους ε, πολίτες της χώρας, του βασιλείου, αλλά ο τρίτος ήταν σοφός και ήξερε ότι με το αλάτι και τη ζάχαρη η ζωή σου γίνεται καλύτερη. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάθε σου γεύμα. Ε, και νομίζω ότι ακριβώς το αλάτι και τη ζάχαρη είμαστε εμεί ω Επιτροπή σε σχέση με το Κοινοβούλιο και αυτό κάνει και τη διαφορά. Έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα. Τούτου λεχθέντος, σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας και έχω να αναφέρω αρκετά πράγματα. Πρώτον, η έκθεση αυτή είναι οριζόντια Γι' αυτό θέλω, επειδή πρέπει να είμαστε συνοπτικοί, να αναφέρουμε. Ε, Καταρχά, την ανάγκη οι εκτελεστικοί οργανισμοί να χρησιμοποιούν καινού διαγωνισμού για να υπάρχει θεματική διασύνδεση ανάλογα με του ε, τομεί αρμοδιότητα και για να υπάρχει και εναρμόνιση. Ενώ ότι κάποιοι εκτελεστικοί οργανισμοί μπορεί να έχουν πολύ κοινέ ανάγκε ό,τι αφορούν ε, τι δημόσιε προμήθειε. Άρα μπορούν να ενώσουν τι προσπάθειέ του ε, για να ε, υπάρξει εναρμόνιση και τυποποίηση και να υπάρχουν κοινοί κανόνε. Ε, αυτό θα βοηθήσει όσους ε, υποβάλλουν προσφορές ε, σε ένα δημόσιο διαγωνισμό και σίγουρα θα οδηγήσει σε απλούστευση τη όλη κατάσταση για του εκτελεστικού οργανισμού που έχουν παρόμοιε, για να μην πω ίδιε ανάγκε, για την συντήρηση ε, των οχημάτων, για τη συντήρηση των κτηρίων. Νομίζω θα μπορούσαν με εναρμονισμένο τρόπο να προχωρούν για την ε, δημοσίευση διαγωνισμού. Έχω ένα πρόβλημα για τις έδρες. Εμεί έχουμε τρει έδρε. Το να πούμε ότι δημιουργεί δημιουργία αποτελεσματικότητα στο έργο των οργανισμών, το ότι μπορεί να έχουν παραπάνω από μια έδρα, θα μπορούσαμε να τι χρησιμοποιήσουμε, τις, ε, ε, να τα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα, επειδή έχουν μια έδρα. Επίση, διερεύνηση νέων πηγών χρηματοδότηση. γιατί έχουμε το Brexit. Και θα επηρεάσει αυτό τις ε, άμεσες συνεισφορές προς κάποιους οργανισμούς. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της έλλειψης ικανοποίησης, γιατί ζητάμε συνέχεια από του οργανισμούς να κάνουν περισσότερα με λιγότερους σπόρους και λιγότερο προσωπικό και καταλαβαίνω πώς νιώθουν. Ζητάμε όλο και περισσότερα από τη διοίκηση. Όλο και περισσότερες ευθύνες και καθήκοντα τους ζητάμε να αναλάβουν, αλλά θέλουμε να παίρνουμε και λιγότερα. Δεν ξέρω αν ένας μαθηματικός ε, υπάρχει στον κόσμο που θα μπορούσε να λύσει αυτή την εξίσωση. Και θα το δούμε και στι διαπραγματεύσει για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ, θα το δούμε και στον προορισμό του 20. Ε, οι δημόσιε προμήθειε είναι άλλη μια αδυναμία, ένα δυνατό σημείο. Για πέντε λόγου. Ε, και θα ήθελα επίση ε, και η αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων και οι μάρτυρε μου συμφέροντο να περιληφθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι μεμονωμένου εκτελεστικού οργανισμού, θα ήθελα να εστιάσω στην ΕΑΣΟ καταρχά, που πράγματι είχε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο, αλλά έκτοτε έχει έναν ε, ενδιάμεσο, είχε έναν προσωρινό και τώρα έχει τον ε, διευθυντή, τη διευθύντρια τη νέα και η πρόοδος είναι θεαματική. Είδα την νέα οργανωτική δομή, ε, σε επαφές που είχα, είδα και κάποια διορθωτικά μέτρα. Το πιο σημαντικό εδώ είναι να γνωρίσουμε την πρόοδο, πιστεύω. που εμένα με έπεισε τα έγραφα που διάβασα ότι υπάρχει. Τώρα, για τον εσωτερικό έλεγχο. Το Σεπτέμβριο του 2019. έχει η Άσο ε, βελτιώσει την οργανωτική διακυβέρνηση και προσπαθεί να δημιουργήσει και την εσωτερική ε, δομή ελέγχου. Το ίδιο συμβαίνει με τον ίδιο Λίσα Frontex. Δύσκολο το 18, ε, δύσκολο και το μεταβατικό έτος το 19. Θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε κυρίως στην πολιτική προσωπικού και το σύστημα εκ των υστέρων επαλήθευσης. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα τώρα, ε, τη ΦΡΑ. Μετά από τις επαφές που είχαμε υπάρχουν κάποια θέματα τεχνικά που πρέπει να διορθωθούν. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης. Υιοθέτησε πρόσφατα εκτελεστικούς κανόνες για την πρόσβαση στα δημόσια για το Οργανισμό Χημικών Ουσιών η εξπόστα παλήθευση με ενδιαφέρει. Το είπαμε και στην ακρόασή μας το Δεκέμβριο. Με αυτά θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά αρνητικά, το πει το Brexit, την έλλειψη προόδου, τουλάχιστον να κάνουμε κάτι θετικό με τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Και ξέρω ότι είναι εύκολο ε, να μιλάμε εδώ ε, από θέση ισχύω ε, και να καλούμε τους διευθυντές να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να πάμε και εκεί για να δούμε τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για τους οργανισμούς και την απαλλαγή για το 2018. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Θα δώσω το λόγο στη Λάρα Βόλτες ω σκιώδη συγκήτρια για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια οριζόντια σχόλια πρώτα και ύστερα θα μπω σε λεπτομέρειες ε, με κίνδυνο να πω τα ίδια με τους ε, προλελήσαντε. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ του ε, τους για την έκθεση που συνέταξαν για τους 30 33 οργανισμούς, 33 υπηρεσίες. Δεν ήταν εύκολο σίγουρα ούτε για εσάς ούτε για τους και οδησηγητές. Τώρα θα ήθελα να κάνω τρία οριζόντια σχόλια. Το πρώτο αφορά την ίση εκπροσώπηση των φύλων. Αυτή τη στιγμή στην έκθεση δεν υπάρχει κάποιο κεφάλαιο για ε, την ίση εκπροσώπηση των φύλων στις υπηρεσίες αυτές, κάτι που υπήρχε στην έκθεση του 2017 και είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να συμπεριληφθεί. Θα καταθέσω λοιπόν τροπολογίες σχετικά. Σε ό,τι αφορά την, ε, τις εκθέσεις για την βιωσιμότητα, να σας υπενθυμίσω ότι το ελεκτικό συνέδριο δημοσίευσε μία έκθεση σύμφωνα με την οποία παρά το ότι οι περισσότερες υπηρεσίες δίνουν λεπτομέρειες για θέματα βιωσιμότητας, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τη διαχείριση, για παράδειγμα, των πλαστικών απορριμμάτων, για τις επιπτώσεις που ε, αυτό έχει εξωτερικά ως προς τη βιωσιμότητα και θα ήθελα να αναφερθεί και αυτό στην έκθεση. Τέλος, να προσθέσω κάτι για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας των ε, έκτακτων υπαλλήλων, κάτι το οποίο χρειάζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες. Και τώρα, πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την ΕΑΣΟ, υποστηρίζω τα θετικά σχόλια, χρειάζονται όμως αρκετές ε, τροποποιήσεις έτσι ώστε να λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και τις παρατυπίες ε, των ε, πληρωμών της ΕΑΣΟ για το έτος 2018. Επίσης, θα έπρεπε ίσως να συμπεριλάβουμε κάποιες συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, για παράδειγμα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί ο συντονισμός με τις άλλες υπηρεσίες και για τα συμπληρωματικά μέτρα. Ε, τέλος να πω ότι μας χαροποιεί το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στην ΕΑΣΟ. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Να τονίσω καταρχάς ότι πρέπει να αποφύγουμε ε, συγκρούσεις συμφερόντων μετά τη λήξη μιας ε, σύμβασης εργασίας εκεί. Ήδη στην Ολομέλεια της περασμένης εβδομάδας ε, συζητήσαμε το θέμα του κύριου Φάρκας, ο οποίος ήταν μέλος της ρυθμιστικής αρχής της ε, ΕΤΑ και τώρα έχει βρει απασχόληση σε ένα λόμπι, ομάδα ασκήσης πίεσης. Ζητήσαμε λοιπόν από τους ευρωβουλευτές να μην ε, συναντηθούν με τον κύριο Φάρκας και θα ήθελα να συμπεριληφθεί και αυτό στην έκθεση. Σε ό,τι αφορά ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. Την τελευταία φορά που βρέθηκα εκεί διαπίστωσα ότι υπήρχε πρόβλημα με την ε, συλλογή των ε, οικονομικών εισφορών, των τελών, το οποίο αποτελούσε το 73% των πόρων της υπηρεσίας αυτής. Η συλλογή όμως των τελών αυτών εξαρτάται απόλυτα από τις ε, δηλώσεις των όσων πρέπει να καταβάλουν εισφορές, επιχειρήσεων κτλ. Και έχουμε εδώ περιπτώσεις ε, που έχουν σημειωθεί παρατυπίες, ε, επιχειρήσεις που λένε πως είναι πιο μικρές από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό επηρεάζει την, τις εισφορές που πρέπει να καταβάλουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. Και έτσι αναμένεται το 2019 να μειωθούν τα έσοδα τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε κάποια λύση για να καλυφθούν οι απώλειες. Τέλος, ε, σε... Το ελεκτικό συνέδριο έχει επιστήσει την προσοχή σε θέματα ε, συμβάσεων για υπαλλήλους πληροφορικής. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάρα. Η κυρία Στουκάρδιου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές. Θα ήθελα με τη σειρά μου να εστιάσω σε κάποια γενικότερα θέματα. και κάποια συστημικά προβλήματα τα οποία θεωρώ πως πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παρότι με χαροποιεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται τα θέματα επιδόσεων, θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες για τον κάθε οργανισμό. Έπειτα, να σημειώσω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και συγκεκριμένη πολιτική για αυτό το θέμα της, ε, του περάσματος από τον ε, δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Πώς μπορούμε δηλαδή να ελέγξουμε το πού θα βρουν απασχόληση οι πρώην υπάλληλοι αυτών των ε, φορέων. Χρειάζονται σίγουρα καλύτερη έλεγχη, σαφέστεροι κανόνες. Σε ό,τι αφορά τους ε, μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος, υπάρχουν μεν κανόνες, όμως σε καμία από αυτές τις υπηρεσίες δεν έχει παρατηρηθεί κάποια περίπτωση σχετική σε κανέναν από, αυτούς, του, από αυτές τις, ε, σε καμία από αυτές τις υπηρεσίες, ούτε τα θεσμικά όργανα. Αυτό τι σημαίνει, είτε ότι το προσωπικό δεν έχει επίγνωση των κανόνων, είτε ότι δεν εμπιστεύεται το σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν νομίζω πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πουθενά. Ωραίο θα ήταν, αλλά είναι απίθανο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται λοιπόν να αυξήσουμε την ε, ενημέρωση, να ευαισθητοποιηθούν οι υπάλληλοι, να διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι έτσι ώστε να βοηθήσουμε ε, όσους καταγγέλουν παρατυπίες να αποκαλύπτουν τις ε, πληροφορίες ε, αυτές για τις περιπτώσεις όπου βλάπτονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, από τη μία υπάρχει διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντική, οι θεσμοί και οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα, να λειτουργούν υποδειγματικά και να ξεπερνούν ε, τα όσα προβλέπει το νομικό τους πλαίσιο. Όλοι θα έπρεπε να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις εμβάσεις που χορηγούνται και ε, όχι μόνο για, για ποσά πάνω από 15.000 ευρώ, αλλά και για τα ποσά κάτω από αυτό το όριο. Μετά, ε, διαφάνεια για σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ υπάρχει ακόμα ένα ανεπίλητο πρόβλημα παρά τις βελτιώσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ λοιπόν πως έχει έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα κοινό ενωπημένο μοντέλο έτσι ώστε να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων ε, και με τον τρόπο αυτό να αποφύγουμε ορισμένα πρώην μέλη διοικητικών συμβουλίων να λένε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, δεν υπάρχει συγκρούση συμφερόντων στη νέα μου δουλειά. Ψηφιοποίηση. Εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία οι υπηρεσίες αυτές να αυξήσουν την ε, διαφάνεια και την λογοδοσία. Χρειάζεται να ε, ενισχύσουμε την ψηφιοποίηση και να γίνει αυτό ταχύτερα καθώς και να εφαρμοστεί με τον σωστό τρόπο ε, οι διαγωνισμοί και η ανάθεση συμβάσεων θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά και αυτό θα βοηθούσε σε όλους αυτούς τους τομείς που προανέφερα. Σε συνέχεια του θέματος των δημοσίων συμβάσεων, δυστυχώς έχουν εντοπιστεί κάποια συστημικά προβλήματα. Ορισμένες υπηρεσίες, ε, για παράδειγμα, έχουν προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά τα, τις ε, συμβάσεις ε, για θέματα πληροφορικής. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα πληρωμών ακριβώς λόγω της λάθος χρήσης, των, λάθος εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Χρειάζονται όχι μόνο σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και επαρκής κατάρτιση για το προσωπικό. Έπειτα, στελέχωση υπηρεσιών, Ορισμένε υπηρεσίε είναι πιο ελκυστικέ από κάποιες άλλες. Ε, αυτό το άκουσα στο πλαίσιο τη συζήτηση για τι προσλήψει, ότι ορισμένε υπηρεσίε αντιμετωπίζουν πρόβλημα να βρουν ανθρώπινο δυναμικό. Ε, η στελέχωση μια υπηρεσία είναι και αποτέλεσμα καλού μάρκετινγκ μεταξύ άλλων. Θα μπορούσαμε ίσω να δούμε ε, πώ θα χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά μέτρα, όπω για παράδειγμα βοήθεια προ την οικογένεια, μισθολογική αντιστάθμιση, ενίσχυση, θα πρέπει να δούμε όλες τις συνιστώσεις που μπορούν να κάνουν μια υπηρεσία πιο ελκυστική. Για παράδειγμα, ε, μπορούμε να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα ορισμένων υπηρεσιών που έχουν ε, συνοδεύσει την ε, υπηρεσία από ένα ευρωπαϊκό σχολείο, έτσι ώστε να μπορούν πάλι να στείλουν τα παιδιά τους εκεί. Τέλος, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαλλαγή με το σύστημα νη συνένα για φέτο. και θα ολοκληρώσω λέγοντα ότι σα ευχαριστώ όλου για τη σκληρή δουλειά σα. Η ομάδα μα φυσικά θα καταθέσει τροπολογίε και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία με όλου σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. base out από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και τους τρεις συνεισηγητές και ελπίζω ότι ο ασθενής που απουσιάζει σήμερα θα γίνει σύντομα καλά. Σας ευχαριστώ πάντω και τους τρεις, καθώς επίσης και τη Γραμματεία και όλο το προσωπικό της Επιτροπής μας που σας επέτρεψε να καταρτήσετε τις σημαντικότατες αυτές εκθέσεις και να επιτελέσετε το σημαντικότατο αυτό έργο. Η βάση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή για τη δική μας την ανάλυση είναι πολύ θετική και μας επιτρέπει να καταθέσουμε και πιο εξειδικευμένες ε, τροπολογίε. Να καταφέρουμε και εμεί να προσθέσουμε, να το θέσω έτσι, τη ζάχαρη και το αλάτι στην έκθεση αυτή. Και κάνω τη μια αφορά σε αυτό που είπε ο κύριο Νάβοκοφ πριν από λίγο. Καταρχάς, ε, συμφωνούμε με τον προλύσαντα από την ομάδα των σοσιαλιστών ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με τους έκτακτους προσωρινά απασχολούμενους με την ανάθεση συμβάσεων. Θα πρέπει προφανώς οι πτυχές αυτές να καλύπτονται πλήρως. Το είπε και ο συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σαφώς υπάρχει ένα πρόβλημα με την κατανομή των κονδυλίων προς τους οργανισμούς αυτούς. Οργανισμοί οι οποίοι λαμβάνουν όλο και λιγότερα χρήματα, μόλον ότι αυξάνονται οι αρμοδιότητε και ευθύνε του. Και αυτό το είδαμε περίτρανα με την περίπτωση τη Ευρωπαϊκή υπηρεσίες υποστήριξη για το άσυλο με την ΑΖΟ, αλλά δυστυχώς ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουμε και σε άλλους οργανισμούς, ιδίως με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα όσον αφορά τις διαπραγματεύσει για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν δούμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως, φαίνεται ότι ένα τεράστιο έργο θα αναλυφθεί αυτή τη φορά από τους εξωτερικούς οργανισμούς Τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν την απαραίτητη στελέχωση καθώς επίσης και τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους. Ως προς αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μολονότι το είχαμε τονίσει αυτό και σε προηγούμενες απαλλαγές. Όσον αφορά τώρα την ΕΑΣΟ. Προφανώ έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδο. υπάρχει βελτίωση, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επικρίνουμε τον οργανισμό αυτό διότι από ό,τι φαίνεται είναι τεράστιες οι πολιτικές απαιτήσεις και προσδοκίες από αυτόν τον οργανισμό και από την άλλη φαίνεται ότι ο προπολογισμό που έχει δοθεί στον οργανισμό αυτό δεν το επιτρέπει να αποκριθεί στι προσδοκίε αυτέ. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Σε αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε και όχι τόσο πολύ σε ποιον θα καταρρύψουμε τελικά τι ευθύνε. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και με τον Frontex. Ανάλογε τάσει και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό περιλαμβάνει βέβαια και το προσωπικό του οργανισμού. Ιδίω για τους ανθρώπους αυτούς που εργάζονται στην ακτοφυλακή και στην οριοφυλακή. Θα υποβάλουμε και σχετικές τροπολογίες όπως έγινε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τώρα για τους υπόλοιπους οργανισμούς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επικεντρωθούμε στη σύγκρουση συμφερόντων. Ως συνήθως, κοιτώντα καταρχάς την ΕΦΣΑ, βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν ε, εκεί συγκεκριμένοι κανόνες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 25%. Καταλαβαίνετε ότι είναι υψηλό ενδεχομένω το ποσοστό αυτό. Θέλουμε πραγματικά να τηρήσουμε την ανεξαρτησία που θα πρέπει να έχει ο οργανισμός αυτός και ξέρετε ότι και για την, τον οργανισμό φαρμακευτικών προϊόντων έχουμε ένα αντίστοιχο ποσοστό 90%. Καταλαβαίνετε ότι και με τον οργανισμό αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε, καθότι έχει πάρα πολλέ επαφές με τον ιδιωτικό τομέα και μπορεί ενδεχομένω να έχουμε προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, το ζήτημα της μετάβασης από τον δημόσιο στο ιδιωτικό τομέα το είπε και αυτό ο συνάδελφο από την ομάδα Renew, έχουμε εγκρίνει ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η διατύπωση που έχουμε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ πιο αυστηρή από τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο σημείο τη έκθεση αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αυστηρότη διατύπωση με την οποία έχουμε επικρίνει τη μετάβαση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, στα πλαίσια τη CBA πάντα, ακολουθούνται κάποιοι νέοι κανόνε όσον αφορά την καταπολέμηση τη νομοποίηση παράνομων εσόδων και εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αυστηρή διατύπωση που έχουμε εγκρίνει σε άλλα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει και εδώ να γίνεται μια αντίστοιχη μνήα. Όσον αφορά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όντως έχουμε μερικές περιπτώσεις όπου τα πράγματα δεν κινήθηκαν πολύ σωστά. Συμφωνώ λοιπόν με τον συνάδελφο από το Renew ότι θα πρέπει οι κανόνες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύουν για όλους τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στους οργανισμούς αυτούς. Είναι πολύ περίεργο να έχουμε τόσα λίγα περιστατικά όπου δραστηριοποιούνται τελικά μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Μήπως τελικά δεν μπορούν να αναλάβουν ελεύθερα δράση, μήπως δεν του έχουμε δώσει τα απαραίτητα κίνητρα για να δραστηριοποιηθούν θα πρέπει έπειτα να ακολουθήσουμε και τις συστάσεις που έκανε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια όσον αφορά τους εξωτερικούς αυτούς οργανισμούς και άλλωστε ρόλος μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην έμπρακτη εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Τέλος. Μετακινήθηκαν δύο οργανισμοί, η EMA και η EBA, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα οι ελεγκτέ από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να κάνουν και έναν έλεγχο για να μα πούνε τελικά αν όντω ακολουθήθηκαν βέλτιστε πρακτικέ κατά τη μετακόμιση των δύο αυτών οργανισμών εκτό Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει όντω εδώ πέρα να δούμε ότι τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά συμπληρώνοντας αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Λεκό Κόμμα και από το Renew Europe και νομίζω ότι και με τις τροπολογίες που θα καταφέρουμε να καταθέσουμε θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε ένα σύνολο πολύ θετικών εκθέσεων προκειμένου πραγματικά να επιφέρουμε και εμείς το αλάτι και τη ζάχαρή μας στην όλη αυτή τη διαδικασία. Ο κύριο Ντεχόφσκι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή φαίνεται ότι αρεσκόμαθα να ακούμε ή να λέμε ιστορίε, εδώ να σα διηγηθώ κι εγώ μια ιστορία. Μια ιστορία που μου είχε διηγηθεί ο πατέρα μου όταν ήμουν παιδί για μια πριγκίπισσα που έπρεπε να διαλέξει τον ε, σύζυγο ε, και ήταν πάρα πολύ ε, όμορφος ο πρώτος υποψήφιος ο δεύτερος ήταν πάμπλουτος ε, και είχε πάρα πολύ μεγάλη έτσι, υπόλοιψη. Και ο τρίτος υποψήφιος ε, είχε ένα καθρέφτη στο χέρι του και της είπε «Κοιτάξτε ο καθρέφτη». Ε, ποια ήταν η επιλογή της πριγκίπισσας. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν επελέγει ο πρώτος ή ο δεύτερος, ε, δεν θα ήταν ε, αυτή η πριγκίπισσα μέλος αυτής της Επιτροπής. Ο πρώτος και ο δεύτερος υποψήφιος δεν έχουν θέση ε, στην δική μας την Επιτροπή. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τον καθρέφτη, αν θέλουμε λοιπόν την αλήθεια. Η πριγκίπισσα ήταν έξυπνη. Ήταν έξυπνη, θέλω να ξέρει την αλήθεια και διάλεξε το σωστό γαμπρό τραπεί το Δεν πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να ανησυχούμε τόσο πολύ για το πρόβλημα της ε, εκπροσώπησης των και γυναικών. Έχουμε και άλλα θέματα. Κάποιος μίλησε για το αλάτι και τη ζάχαρη που λείπουν. Να σας πω και εγώ γιατί το λέω αυτό. Υπάρχει έλλειψη πόρων σε πολλούς εκτελεστικούς οργανισμούς. Ε, πολλοί έχουν αναδιαρθρωθεί, έχουν περικοπεί έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή, ε, άλλοι ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και είναι σε κενό ε, και δεν έχουν ε, καμία ιδέα για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον και τι θα τους συμβεί, αν θα καταργηθούν ή όχι. Το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι κανένας δεν διαβάζει ούτε ασχολείται ε, με τα αποτελέσματα του έργου τους. Πλην τη ΕΑΖΟ βέβαια. Υπάρχουν αιτήσιε εκθέσει από πολλού εκτελεστικού οργανισμού, αλλά δεν του δίνει καμιά σημασία αυτών των εκθέσεων και δεν τι διαβάζει κανένα. Και πολλοί εκτελεστικοί οργανισμοί από τότε που ιδρύθηκαν έχουν χάσει το λόγο ύπαρξή του πια. Μπορεί να ε, σκεφτεί κάποιοι το Δουβλίνο ή την Ελλάδα, αλλά εγώ μιλάω γενικά. Μήπως πρέπει να κρατήσουμε τον καθρέφτη και να κοιταχτούμε να πούμε έχουμε 34 εκτελεστικούς που τους χρειαζόμαστε. Όχι, δεν τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς. 29 θα αρκούσαν. Ίσως κάποιους θα μπορούσαμε να το συγχωνεύσουμε και να έχουμε ένα πιο ισχυρό οργανισμό στη θέση άλλων ε, περισσότερων. Είχα την ε, τιμή να έχω διατελέσει σκιώδης εισηγητής πολλές φορές για εκτελεστικούς οργανισμούς και είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ όλους σχεδόν τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Αν δεν κοιτάξουμε τώρα όμως τον καθρέφτη, δεν θα δούμε και τι έργο επιτελούν αυτοί οι οργανισμικά, ποιοι έχουν ψηφιοποιηθεί, έχουν, δια... έχουν συρρυκνωθεί σε μέγεθος, έχουν απολύσει κάποιους, έχουν ε, προβεί σε εξορθολογισμό. Τι όμως δεν έχει γίνει και ιδίως από την Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για το ότι παρόλα αυτά δεν χρειαζόμαστε πολλούς από αυτούς τους εκτελεστικούς οργανισμούς και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να είναι και ένας από τους στόχους της διαδικασίας απαλλαγής. Έχει ζητήσει και η Λάρα το λόγο ως απάντηση σε αυτά που είπατε. Ναι, ναι, ζήτησα το λόγο για να πω ότι όσο και αν εκτιμώ αυτές τις ιστορίες, τα παραμύθια που διηγείστε, θα ήθελα να σας ζητήσω να τα εξυγχρονίσετε κάπως, να τα φέρετε στον 21ο αιώνα και να ε, σταματήσουμε αυτά με τις πριγκίπισσες που πρέπει να τις διαλέξει ένας πρίγκιπας. Ε, νομίζω πως δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τέτοια στερεότυπα. Οι πριγκίπισσες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν χρειάζεται να περιμένω τις διαλέξει ο πρίγκιπας. Έπειτα, το παράδειγμα της μιας πριγκίπισσας ε, που ήταν η λίστρια, της άλλης που ήταν ματαιόδοξη, ε, ούτε κι αυτό μ' αρέσει. Έτσι, μια ευγενική υπενθύμηση, έτσι, να τα εξυγχρονίσουμε λίγο αυτά. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό με τις πριγκίπιζες ξέρετε ότι δεν πιάνει ούτε στη Μεγάλη Βρετανία, ούτε στον 21ο αιώνα. Αλλά εντάξει, ιστορίες είναι ιστορίες. Ένα μικρό σχόλιο θα θέλατε να κάνετε, να απαντήσετε. Ναι, καταλαβαίνω ότι κάποιες γυναίκες δεν καταλαβαίνουν την ιστορία αυτή. Προσοχή, προσοχή, λέει η πρόεδρος. Προσέξτε τι θα πείτε. Καταλαβαίνω ε, ότι δεν το καταλαβαίνουν, διότι έχει να κάνει με ιστορία, ιστορικό γεγονός της ιστορίας. Χρησιμοποιώ λοιπόν ένα ιστορικό παράδειγμα για να, να σας εξηγήσω ότι κάποιος έχει προσδοκίες μόνο και μόνο επειδή έχει γεννηθεί σε μια θέση. Δεν έχει να κάνει με πρίγκιπες και πριγκίπισες, έχει να κάνει με τον καθρέφτη που πρέπει να ε, έχουμε, να κοιταχτούμε για να δούμε την αλήθεια. Αυτό είναι το ζουμί της ιστορίας. και αν δεν θεωρείτε έξυπνη την ιστορία, εντάξει δεν χρειάζεται να είναι πάντα έξυπνη μια ιστορία και αν τη μεταφέρουμε στον 21ο αιώνα μπορεί ίσω ξέρετε, να μην καταλάβει κανείς ε, τι θέλουμε να πούμε. Η ιστορία αυτή είναι ένας καθρέφτης και μας λέει τι χρειαζόμαστε εμείς σαν ε, ευρωπαϊκός θεσμός. Ωραία. Ωραία. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε και με τα παραμυθάκια, τις ιστορίες. Φτάσαμε στο τέλος της ε, συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Τέσσερα πολύ μικρά σχόλια έχω να κάνω πρωτού κλείσουμε για σήμερα. Νομίζω πως ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ε, υπηρεσιών αυτών. Τι δυνατότητες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει, ποιο είναι τα μέλη των ε, διοικητικών συμβουλίων αυτών των οργανισμών, ποιες είναι οι δυνατότητες επίβλεψης και ελέγχου που έχει η Κομισιόν. Η Κομισιόν θα πρέπει να έχει εποπτικό ρόλο και θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο λοιπόν με αυτό. Έπειτα, αυτά που είπε ο συνάδελφος για την ε, συνιστόσα διόρθωσης, ε, ναι, έχει δίκιο. Θα χρειαστεί να υπάρξει μια καλή, ε, ένας καλός συνδυασμός από όλα τα κράτη-μέλη και τα 27 ακριβώς λόγω αυτού του συντελεστή διόρθωσης. Ο κύριος Έικουτ επίσης έκανε μία ερώτηση για ε, την ταχύτητα των εξελίξεων, των ε, ανακοινήσεων, των αναδιαρθρώσεων σε μία επιχείρηση. Δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε πρέπει να αλλάξει η δομή ορισμένων υπηρεσιών, να βελτιωθεί. Η Frontex είναι μια υπηρεσία για την οποία έχουμε συζητήσει αρκετά, αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε μήπως μπορούμε να ε, κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς και να ομοδοποιήσουμε κάποιες ανάγκες. Τώρα, έχει προκύψει και κάτι άλλο πιο πολύπλοκο. Όταν υπάρχει ένας ε, ειδικό σε έναν τομέα, είτε αυτό είναι περιβάλλον, είτε αυτό είναι χημικά, α πούμε, οτιδήποτε άλλο. Τι θα κάνουμε όταν τελειώνει η σύμβασή του για να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Είτε θα συνεχίσουμε να τον πληρώνουμε, για παράδειγμα, για τα δύο επόμενα χρόνια, για να μην βρει απασχόληση αλλού και προκύψει θέμα σύγκρουση συμφερόντων, ή θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το κάνουμε, διότι δεν μπορεί κάποιος ε, ειδικό να προσληφθεί με διετή, ας πούμε, σύμβαση και μετά εμείς να περιμένουμε να ε, είναι, έχει έμυθος και να τηρήσει σιωπή για τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο ερώτημα αυτό. Και μάλιστα με αφορμή την περίπτωση του κύριου Φάρκα ε, το σκέφτηκα πολύ. Και σίγουρα ένας ειδικό σε τραπεζικά θέματα δεν μπορεί να πάει να βρει δουλειά σε έναν οργανισμό χημικών, α πούμε, διότι δεν είναι ε, το πεδίο του αυτό. Γι' αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτά τα, αυτές οι διετής ή πενταετής συμβάσεις είναι ο σωστός ε, τρόπος απασχόλησης, αν έχει νόημα να τους δίνουμε τέτοιες συμβάσεις ή αν πρέπει να αλλάξει αυτό. Αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί ακόμα ε, και σε περιπτώσεις απασχόλησης στο περιβάλλον ε, και σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η Food Watch, ας πούμε, δεν είναι μία απλή ΜΚΟ, είναι ένας ολόκληρος όμιλος. Και φέρει τη δική του προστιθέμενη αξία όπου παρεμβαίνει. Και πιστεύω ότι το θέμα αυτό ε, συνδέεται άρρηκτα με ε, οικονομικές επιπτώσεις. Βέβαια, δεν μπορούμε να απασχολήσουμε πάρα πολύ τις ε, αντίστοιχες επιτροπές περιβάλλοντος και οικονομικών, όμως ε, θέλει μεγάλη προσοχή και να εξετάσουμε όλες τις ε, συνέπειες. Τώρα, ένα λεπτό ακόμα για το ελεκτικό συνέδριο και δύο άλλα πράγματα ακόμα. Μπας, ας μην χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια για να καλυφθούν οι ελλείψεις ε, στις ε, εισφορές που πρέπει να πληρώσουν στις υπηρεσίες αυτές. Ε, εδώ δεν μπορούμε να σκίσουμε πίεση όσο και να το θέλαμε. σε ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να διαπιστώσουν κάποια πράγματα, όμως δεν μπορούν να παρέμβουν. Όταν κάποιος πληρώνει εισφορές, εγώ δεν έχω πρόβλημα, σωστά το κάνει. Δεν βλέπω δηλαδή κάποια ε, δυσκολία ή κάποια περίπτωση που μπορεί να ασκήσει επιρροή μια ε, επιχείρηση που πληρώνει εισφορές σε έναν ε, οργανισμό, είτε είναι φαρμακευτική, είτε οτιδήποτε άλλο. Διότι στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, εγώ γνωρίζω ότι με τις δικές μου εισφορές θα καλυφθούν τα έξοδα, τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας. Δεν μπορώ όμως να επηρεάσω την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων για ένα φάρμακο ή μπορώ. Σε περίπτωση που επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ένα προϊόν, εκεί έχω πρόβλημα. Αλλά αυτό φοβάμαι πως θέλει πιο εντατική συζήτηση. Θα δώσω όμως ένα τέλος στο σημείο αυτό. Τελειώσαν τα παραμυθάκια και ιστορίες για σήμερα. Θα συναντηθούμε ξανά στις 2.30 το μεσημέρι. Δυστυχώς, ε, ξέχασα να αναφέρω την καταληκτική ημερομηνία για τις ε, εκθέσεις ε, και θα σας πω ότι πρέπει να το κοιτάξετε, να προσέξετε την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης λογιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι εισηγητές θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πριν τελειώσουμε. Όλα εντάξει. Ναι, όλα, όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τα ξαναλέμε στις 2.30.